Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε θερμά στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής το νέο έτος 2011. Εύχομαι σε όλους ένα υγιές έτος και γεμάτο επιτυχίες για τις διάφορες, ε, τα διάφορα εγχειρήματα που έχουμε υπό ανάπτυξη και φυσικά κάθε επιτυχία στη δουλειά της ε, Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Και πιθανότατα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι και πάλι θα είναι μια πολυσχηδής, ένα πολυσχηδές εύρος θέματων, θεμάτων, με συγχωρείτε, όπως ε, πάντα ήθιστε. Και ξεκινάμε καλά, με καλό τρόπο. Έχουμε πλούσια ημερήσια διάταξη, ήδη σήμερα κιόλας. Και η γραμματεία ήδη μου έδωσε μια προειδοποίηση να μην υπάρχουν παρεμβάσεις πάνω από δύο λεπτά για να τα καταφέρουμε από πλευράς χρόνου διότι θα έχουμε και πολλές ψηφοφορίες που θα διεξαχθούν αύριο. Και έτσι στο μεγάλο βαθμό θα πρέπει να μπορέσουμε να ε, επεξεργαστούμε αυτά τα θέματα πριν από τις ψηφοφορίες σήμερα. Χαιρετίζω λοιπόν όλους και εύχομαι κάθε επιτυχία στη δουλειά μας να συνεργαστούμε με θετικό τρόπο και σε όλα τα θέματα να σημειώσουμε πρόοδο επί της ουσίας. Και περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει μια μικρή τροποποίηση. Είχαμε διαβάσει στις ειδήσει ότι το σύστημα εμπορίας ρήπων και πάλι υπέστη επιθέσεις από hacker του κυβερνοχώρου και εγκληματίες αν επιθυμείτε. Και ήταν επιθυμία μας να μας δώσει πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Γενικό Διευθυντής από την Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι με τους συνεργάτες του παρόν και παρόντες όλοι τους ώστε μέσα στο πλαίσιο του σημείου 3 ή δύο ανακοινώσεις του Προέδρου να έχουμε μια σύντομη συζήτηση που θα κάνουμε. Αυτό καθορίζεται και από το χρονοδιάγραμμα κατά τα άλλα. Λοιπόν, παραμένει η ημερήσια διάταξη μετά από αυτή την αλλαγή ως έχει και έτσι εγκρίνεται υποθέτω. Ωραία. Ανακοινώσεις του Προέδρου λοιπόν. Δύο κατηγορίες, δύο ομάδες. Δύο ε, ομάδες θα έρθουν στην ε, Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή αφενός από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Γεωργίας. Σήμερα το απόγευμα θα προσέλθουν και από την άλλη πλευρά θα έχουμε την Οικονομική και ε, Κοινωνική Επιτροπή της Κεντρικής Αφρικής, μια ομάδα που θα παραστεί για να παρακολουθήσει τις ε, διεργασίες και συζητήσεις. Για το άλλο σημείο που προανέφερα, σύστημα εμπορίας ε, ρήπων, ένα κύριο στοιχείο της στρατηγικής μας για την προστασία του περιβάλλοντος, πάλι υπέστη κάποιες επικρίσεις και επιθέσεις εκ νέου. Και αυτό καταδεικνύει ότι αυτό το σύστημα δεν είναι απόλυτα ε, ολοκληρωμένο και στεγανό και υπάρχουν ελλείψεις και έχει προχωρήσει σε σχέση με την εμπορία ρήπων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την Τετάρτη θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι βρίσκεται πίσω από αυτές τις ε, αδυναμίες και ελλείψεις ε, που διαπιστώνονται και έτσι να μην παρακολουθεί και υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα ε, εμπορίας τρύπων. Θα δώσω τον λόγο στο Γενικό Διευθυντή να μας ενημερώσει περί τίνος πρόκειται. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω όλους θα ήθελα να μοιράσω την παρουσίασή μου σε τρία στοιχεία. Πού βρισκόμαστε σήμερα, ποιες είναι οι δράσεις οι οποίες αναλήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα και ποια είναι τα επόμενα βήματα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πρώτον τα γεγονότα. Σήμερα έχουμε μια οδηγία, την ETS, και ξεκίνησαμε από το 2005 να λειτουργούμε σε εκείνη τη φάση υπήρξε μια διαμοιρασμένη ευθύνη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη συνεπώς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουν ε, την ασφάλεια του μητρώου τους. Έχουμε 27 χώρες, έχουμε 27 μητρώα και ακόμα και αν θα πρέπει να πάρουν οι ίδιες οι χώρες τα δικά τους μέτρα, το σύνολο σύστημα θα έλεγα επηρεάζεται από τον ασθενέστερο κρίκο. Αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν ότι από την αρχή του χρόνου έχουμε κυβέρνε... θέσεις υποστή στην Αυστρία, την Ελλάδα και την Τσεχία. Γνωρίζουμε επίσης ότι και άλλα μητρώα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τροτά. Η... Το εύρος της βλάβης δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια. Κάποια εθνικά μητρώα δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως αλλά οι, καλύτερες, ε, οι καλύτεροι υπολογισμοί τους οποίους κάνουμε είναι ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άδειες έχουν μεταφερθεί σε συγκεκριμένους λογαριασμούς σχετικά με τις παραβιάσεις ε, το ασφαλείας και τους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί σε οικονομικό επίπεδο. Αυτά μας οδήγησαν στο να λάβουμε άμεσα προληπτικά μέτρα και η νομοθεσία ETS επιτρέπει ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει την πρόσβαση σε εθνικά μητρώα εάν υπάρχει κίνδυνος για το σύνολο της ασφαλείας των μητρώων και του συστήματος. Ποιες δράσεις αναλάβαμε λοιπόν. Την προηγούμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα διακόψαμε τις συναλλαγές εκτός από τις κατανομές ε, συγκεκριμένου αριθμού συναλλαγών σε όλα τα Μητρώα των κρατών μελών μέχρι την 26η Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα, δηλαδή την Τετάρτη. Τα συζητήσαμε τα θέματα αυτά επίσημα με τα κράτη-μέλη και υπάρχει ομόφωνη υποστήριξη από πλευράς των κρατών μελών για τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να δούμε πώς θα ανατάξουμε την κατάσταση. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διακοπή αφορά τον λεγόμενη αγορά spot μόνο επιτρεπομένων ποσοτήτων και αυτό είναι το μικρό τμήμα της αγοράς άνθρακα, δηλαδή το ένα περίπου πέμπτο ενώ τα περισσότερα γίνονται, οι περισσότερες εναλλαγές γίνονται σε futures και τα futures δεν επηρεάζονται. Λοιπόν, ε, δεν μπορεί κανείς σαν πρόσωπο μεμονωμένα online να κάνει συναλλαγές από τον ένα λογαριασμό στον άλλο, αλλά παρόλα αυτά οι τράπεζες ε, ε, λειτουργούν και μπορεί κανείς να κάνει τις μεταφορές του μέσω των Ιδρυμάτων. Την προηγούμενη Παρασκευή η Επιτροπή Αλλαγής Κλίματος που είναι θα έλεγα το πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε τα θέματα αυτά συμφώνησε με την απέτησή μας ορισμένα ελάχιστα κριτήρια να είναι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των μητρώων και αυτά τα ελάχιστα κριτήρια βασίζονται σε σαφείς αποδείξεις ότι τα εθνικά μητρώα είναι πλέον καταλήλως ασφαλή και έχουν ληφθεί τα μέτρα τα απαιτούμενα για την αντίσταση θα έλεγα σε τέτοιου είδους κυβέρνοεπιθέσεις στο μέλλον. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, σήμερα και αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για τα ελάχιστα κριτήρια, στα πλαίσια των οποίων στα Μητρώα θα επιτραπεί να ξεκινήσουν εκ νέου να συναλλάσσονται. Αυτή τη στιγμή στα ελάχιστα αυτά κριτήρια γίνουν δεκτά από τα Μητρώα, τότε η απαγόρευση λειτουργίας θα αρθεί για το συγκεκριμένο εθνικό Μητρώο. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε ένα προγραμματισμένο ρυθμό επιστροφής σταδιακά από τις προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε γνωρίζουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη <clears throat> έχουν ήδη ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας σχετικά με τα εθνικά τους μητρώα και εφόσον μας αποδείξουν λοιπόν ότι σέβονται τα απαιτούμενα επίπεδα ασφαλείας θα λειτουργήσουν πλήρως συμπερασματικά από το 2012 και πέρα θα υπάρχει ένα συγκεντρωτικό μητρό το οποίο θα το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς τα 27 εθνικά μητρώα των κρατών μελών στην ουσία διακόπτουν την λειτουργία τους από το έτος 2012. Κάποια επιπλέον μέτρα ασφαλείας όπως η διαπίστευση και οι τραπεζικές συναλλαγές online ήδη ε, στην ουσία βρίσκονται εν λειτουργία σε κάποια από τα εθνικά αυτά μητρώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη συστηματικά προετοιμάζει μια τροπολόγηση του κανονισμού λειτουργίας των μητρώων έτσι ώστε να βρεθούν περαιτέρω προϋποθέσεις κοινές για τη την ασφαλή λειτουργία των μητρώων αυτών. Συνεπώς κύριε Πρόεδρε, αυτά έχω να πω προς το παρόν. Υπάρχει μια διακοπή λειτουργίας γιατί όπως είπα έχουμε 27 εθνικά μητρώα, κάτι το οποίο όμως θα πάψει να υπάρχει σαν πρόβλημα από τον Ιανουάριο του 12. Ταυτόχρονα και εν τω μεταξύ θα διασφαλίσουμε το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας για τις συναλλαγές που θα μεσολαβήσουν μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ Διευθυντά για την ενημέρωση. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που υφίσταται επίθεση το σύστημα. Νομίζω προέτους είχε υπάρξει μια υπόθεση απάτης και διαρωτάται κανείς οι χώρες μέλη δεν διδάχθηκαν από αυτά τα συμβάντα ώστε να κάνουν το σύστημα ασφαλές. Πού βρίσκονται τα δύναμα σημεία και ποια μέτρα θα πρέπει να λάβετε ώστε να είναι στεγανό το σύστημα. Σε ορισμένες χώρες, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, σε ορισμένε χώρε είναι ασφαλή τα συστήματα αυτά και σύμφωνα με το παράδειγμα των ασφαλών πρακτικών θα μπορούσε να μεταφερθούν αυτές και σε άλλες χώρες. Τώρα, έχω δύο εγγεγραμμένους. Ο κύριος Φλόρεντς πρώτα. Όταν ακούω τα, για τα θέματα αυτά, αισθάνομαι ομολογώ κάποιο φόβο. Διότι ούτε είμαι σαΐνιστα των υπολογιστών, αλλά μπορώ να φανταστώ κιόλας διάφορες μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω ούτε καν σε ποια χώρα ε, σημειώθηκαν αυτά, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι έχουν δυσκολίες και είναι δύσκολο για μένα να υπερασπιστώ τις αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊ... που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην εκλογική μου περιφέρεια. Και γι' αυτό θέλω να μάθω τι διάθεση συνεργασίας δείχνουν οι χώρες μέλη στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, για ζήτηματα αποβλήτων. Όταν κάπου ανακαλύπτεται καμιά μεγάλη παρανομία, οι χώρες μέλη και οι δικοί μου συμπεριλαμβανόμενοι δεν συνεργάζονται ιδιαίτερα για την αποκάλυψη των προβλημάτων. Ίσως στο τέλος της υπόθεσης, όταν πλέον έχουν αποδειχθεί όλα, για την διόρθωση να είναι πιο συνεργάσιμες. Το σύστημα ITS ε μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα έτσι, διότι το αναμέναμε ότι κάποια στιγμή θα πάθει ζημιά και μπορεί και να καταρρεύσει. Σωστό αυτό, λέει ο πρόεδρος. Chris <coughs> Ευχαριστώ. Ήταν ε, σύντομη η ενημέρωση που μας έγινε, αλλά περιεκτική. Τώρα, υποθέτω ότι πρόκειται για παράνομη, ποινικώς διοκόμενη ε, υπόθεση. Διώκεται κανείς. Ποιος κάνει τις έρευνες, τις ανακρίσεις και προβλέπονται κυρώσεις για αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις. Δεύτερο, ο κύριος Ντεμπέκ είπε ότι η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει μέχρι την 5η, 26 δηλαδή. Ασφαλώς έχει νόημα να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ασφαλές το σύστημα πριν να ξαναρχίσει. Ποιες όμως είναι οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό το trading και η αγορά πόσο θα παραμείνει κλειστή και ποιος καλείται να πληρώσει για όλα αυτά. Ίσως μάλιστα ορισμένα από τα γραφεία αυτά να χρειαστεί να παραμείνουν μόνιμως κλειστά. Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα εάν ένα από αυτά τα registries, από αυτά τα μητρώα μπορεί να αγοράσει κάποιο λογισμικό για να το χρησιμοποιήσει. Και υποτίθεται ότι από το 2012 θα υπάρξει μια κεντρική, ένας κεντρικός οργανισμός. Αυτό θα γίνεται θα παρακολουθείτε από κάποιο ανεξάρτητο οργανισμό ή υπό την ευθύνη των όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις μέσα στην Κομισιόν. Ματίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτά που είπε η Επιτροπή. Είναι μια κλασική περίπτωση αυτών που εμείς ε, συζητάμε υπό την ψηφιακή ημερήσια διάταξη. Θα με ενδιαφέρει από τον, Επίτροπο της, ε, από τον Επιτροπής να ακούσω κατά πόσον σε ευθυγράμμιση με την Έλλη Κρούς που έχει αρκετά πράγματα, 33 νομοθετικά εγχειρήματα, οι προτάσεις πρόκειται να υποβληθούν και για την πολύ σημαντική αυτή αποτυχία είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι υπονομεύεται η εμπιστοσύνη όπως ε, προαναφέρθηκε σε ένα τέτοιο σύστημα και κλονίζεται, κλειδονίζεται η εμπιστοσύνη. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω πόσο εσωτερικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει συντονισμός επ' αυτού. Ξέρω ότι πολλοί εμπλέκονται και συνεργάζονται. Κατά πόσον είσαστε συντονισμένοι ώστε στο μέλλον να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει. Προληπτικά μέτρα να μπορούν να λαμβάνονται ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους συμβάντα. Είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τους πολίτες να λογοδοτούμε εναντί των πολιτών, να μην απολεστεί η εμπιστοσύνη από πλευράς τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ. Κάποιες ε, σύντομες ε, ερωτήσεις ε, για τη ζημιά που έχει σημειωθεί. Και δεύτερον, στο ίδιο σύστημα υπάρχουν ρήτρες ασφαλείας, δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση, για παράδειγμα, τέτοιων διακοιμάσεων θα υπάρχει κάποια δυνατότητα να αποσβεστούν αυτοί οι κλειδονισμοί. Ευχαριστώ. Yeah, das, ich, Πρόεδρος, αυτές ήταν οι ερωτήσεις για το θέμα. Έχετε τον λόγο να απαντήσετε, παρακαλώ. Thank you very much and thank you for the Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι βλέποντας αναδρομικά τα τελευταία αυτά χρόνια, δύο χρόνια, υπήρξαν κάποια τέτοια ολισθήματα ίσονος σημασίας, διαφορετικής φύσεως. Είχαμε και την ιστορία με το ΦΠΑ για παράδειγμα που ήταν ένα γαϊτανάκι για το ΦΠΑ, μπορείτε να δείτε σε σχέση με τα ε, κινητά τηλέφωνα ή τα τσιγάρα κτλ. Αυτά τα οποία είδαμε τις τελευταίες όμως ημέρες ήταν διοργανωμένες ε, οργανωμένες επιθέσεις από κυβερνοεγκληματίες και γι' αυτό άμεσα αναλάβαμε δράση να σταματήσουν οι συναλλαγές ώστε να περιοριστεί η ζημιά. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που είχαν υποστεί επιπτώσεις α, από τέτοιου είδους ίσονος ε, εμβέλειας ε, συμβάντα. Τον Ιανουάριο 2010 γνωρίζουμε ότι η Γερμανία είχε υποστεί μια τέτοια μικρή επίθεση και σε αυτά τα κράτη-μέλη αυτό οδήγησε να αυξηθούν τα επίπεδα ασφάλειας. Κάποια πράγματα έχουν γίνει ήδη λοιπόν και έχουμε ευελπιστούμε ότι πάνω κάτω τα μισά κράτη-μέλη έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Τώρα από την άλλη πλευρά επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάθε συνεδρίαση για τις κλιματικές αλλαγές σε αυτή την Επιτροπή ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να τελούν ενεγρηγόρση, να επιτηρούν την κατάσταση, διότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το οργανωμένο έγκλημα να πλήξει την εμπορία ρήπων. Και αυτά τα οποία είδαμε ως μεμονωμένα γεγονότα τα τελευταία χρόνια διοργανώθηκαν πιο συστηματικά να προσβληθεί το σύστημα με αυτόν τον τρόπο την τελευταία εβδομάδα πρόσφατα. Τώρα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν το πού βρίσκονται εκάστοτε σε αυτό το πλαίσιο και για την δημιουργία αυτού του Μητρώου, αλλά ιδιαίτερα για τα θέματα ασφάλειας ηλεκτρονικής και ψηφιακής ασφάλειας. Αυτά θα πρέπει από τους συναδέλφους όσον αφορά την πληροφορική και την ε, ηλεκτρονική ε, επικοινωνία, IT, συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι μόνο να έχουμε μια καλή επισκόπηση αλλά να έχουμε και τις λύσεις που πρέπει να υιοθετηθούν και να λειτουργήσουν. Πρέπει όμως να τονίσω ότι αυτοί οι hackers στη δραστηριότητά τους έχουν πολύ διαφορετική μορφή στις δράσεις τους. Είναι πολύ επινοητική και πρέπει να δούμε εδώ ότι είναι πολύ οργανωμένη σε αυτή την εγκληματική δράση. Τι γίνεται σε σχέση με τις διακριβώσεις, τις ανακρίσεις. Κυρίως σε εθνικό επίπεδο βρίσκονται, διότι εκεί τα 27 μητρώα βρίσκονται υπό την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους στη διαχείρισή τους. Τούτου λεχθέντος υπάρχουν μεταφορές βέβαια από τη μία χώρα στην άλλη και έχουμε επαφή όχι μόνο με τις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται αυτή την ε, εμπορία, αλλά επίσης και τις εθνικές αρχές, ε, είμαστε σε επαφή με τις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται τους ε, οικονομικούς μηχανισμούς και τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα, διότι αυτό είναι ένα είδους χρηματικής αγοράς, χρηματοοικονομικής αγοράς. Και η Europol έχει εμπλακεί επίσης στην ολοκλήρωση των ανακρίσεων. Αυτές οι διακριβώσεις και ανακρίσεις βρίσκονται ρευστό, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Ένα άλλο θέμα, μια άλλη ερώτηση ήταν ποια, ποιες είναι οι επιπτώσεις, ε, τα συμπεράσματα για τους ε, εμπλεκόμενους στις συναλλαγές αυτές ε, για το άνοιγμα ξανά και για τους 27, τα 27 κρατημέλη. Για να είμαι ειλικρινής δεν αναμένω, δεν προσδοκώ ότι όλα τα 27 μητρώα των εθνικών αρχών θα είναι αρκετά, ας το πω έτσι, ε, υγιή και ε, αποτελεσματικά ώστε να μπορεί να ξαναρχίσει έτσι άμεσα η εμπορία ρήπων. Εξετάζουμε ανακράτως ποιου είδους ασφάλεια, μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί και δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς πόσα κράτη θα είναι έτοιμα εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά δεν αναμένουμε έναν αριθμό που θα είναι πάνω από το ίμιση των κρατών μελών, στο maximum κατά το μέγιστο. Θα ε, έχουμε πάντα μια πολύ προσεκτική επιφυλακτική συντηρητική θέση. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί το θέμα της ασφάλειας από πλευρά κρατών μελών ότι βαίνει καλός δεν θα υπάρξει επανασύνδεση, διότι θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία, την χρηματοοικονομική αξιοπιστία αξιοπιστία αυτής της αγοράς ε, την εμπορία, της εμπορίας ρήπων. Μία εν παρόδο παρατήρηση, δεν έχουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία, κάποια τεκμήρια ότι α, ε, υφίσταται απειλή η ίδια η υγεία ή το πλαίσιο της αξιοπιστίας του συστήματος. Είναι το χρηματοοικονομικό ας το πλαίσιο το οποίο έχει υποστεί πλήγματα. Ετοιμαζόμαστε τώρα για το κεντρικό μητρό. Μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί από έναν εξάρτητο φορέα να αναλάβει αυτό το έργο. Δεν έχουμε ακόμα λάβει αποφάσεις επ' αυτού. Όμως είναι μία από τις εναλλακτικές λύσεις που αυτή τη στιγμή εξετάζουμε στο τρέχον έργο μας. Επίσης υπήρξε μια ερώτηση για τις διακοιμάσεις τιμών και πώς τις αντιμετωπίζουμε στη διαχείριση. Όσον αφορά τις διακοιμάσεις τιμών ήταν σχετικά περιορισμένες πρόσφατα και μάλιστα ήταν σχετικά σταθερή η τιμή του άνθρακα μεταξύ 14 και 16 ευρώ ε, για τον τόνο άνθρακα. Δεν ε, προβλέπουμε κάποια προβλήματα και όμως οι απώλειες όπως ε, εκτιμήθηκαν είναι περίπου του ύψους 2 εκατομμυρίων επί ε, για παράδειγμα 14 τόσα 15 ευρώ για παράδειγμα και θα δείτε την μέγιστη απώλεια που έχουμε υποστεί ή που αξιολογούμε, εκτιμούμε ότι έχει, έχουμε υποστεί έχουμε ε, λάβει και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα και απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη όχι μόνο να δράσουν έτσι αλλά και να ανακτηθούν οι απώλειες ε, που έχουν σημειωθεί από τους ε, οικονομικά εμπλεκόμενους. Και υπό αυτό το πρίσμα αν είναι μικροί ή μεγάλη οικονομικά εμπλεκόμενοι δίνουμε παρόλα αυτά τεράστια σημασία στην ασφάλεια του συστήματος συνολικά. Και θα περάσουμε σε πολύ πιο σκληρές διαπραγματεύσεις και συζητήσεις όσον αφορά τα κράτη-μέλη για να αποφευθεί κάτι τέτοιο όπως αυτό που σημειώθηκε στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό απαντώντας στις ερωτήσεις και τοποθετούμενοι για τα σχόλια που έγιναν. Ευχαριστώ. Επερώτηση, Chris Davis. Implications for the people who are... Τώρα, για όσους αγοράζουν τις αλάουνσες αυτές, έχουν επαρκές περιθώριο για να καλυφθούν μέχρι ότου ξανανοίξει η αγορά. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο, το κεντρικό μητρό να το αναλάβει ένα ειδικό οργανισμός ανεξάρτητος που θα, είναι και, που θα έχει και τα επαρκή μέσα ώστε να, να τον ε, ασφαλίσει, το, να ασφαλίσει το, το Μητρό. Ναι, απάντηση. Ναι, πιθανόν θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη ενός ανεξάρτητου οργανισμού. Ε, ψάχνουμε και τα υπέρ και τα κατά. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει επιληφθεί ένας ειδικό. Δεν είμαι βέβαιος ότι και σε όλες τις χώρες μέλη είναι στο ίδιο επίπεδο γνώσης οι ειδικοί που χειρίζονται τα μητρώα αυτά. 27 διασυνδεμένα μητρώα σημαίνει βέβαια η διαδικτύωση αυτή ότι η ασφάλεια εξαρτάται από το πιο ασθενές μέλος. Τώρα, οι ζημίες μπορούν να διορθωθούν και να επανακτηθούν τα απολεστέντα. Αυτό εξαρτάται από την νομοθεσία που διέπει τα Μητρώα στο εθνικό επίπεδο. Σε ορισμένες χώρες μέλη ανάκτηση των απολεσθέντων, των ζημιών είναι δυνατή. Σε άλλες χώρες μου λένε όχι. Εφόσον δεν είναι εναρμονισμένη εναρμονισμένο το δίκτυο δεν θα έχουμε και ενιαία λύση. Συζητούμε πάντως με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς για να φτιάξουμε μια νομοθεσία για τις αγορές για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε το σύστημα ETS έτσι ώστε να έχουμε την μέγιστη νομική κάλυψη και όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια σύνταξης των νομοθετημάτων αυτών θα σας υποβληθούν. Ελπίζω το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο. Πρόεδρος Λάινεν, τα συμβάντα αυτά δείχνουν τι σημασία έχει, τι μεγάλη σημασία έχει ένα ευρωπαϊκό κεντρικό σύστημα και όχι 27 ξεχωριστά εθνικά συστήματα εμπορίας που στην ουσία προκαλούμε έτσι τους εγκληματίες να ψάξουν να βρουν τα παραθυράκια. Ελπίζω ότι οι ειδικοί που προσλαμβάνετε θα είναι αρκετά ικανοί ώστε να ασφαλίσουν το σύστημα. Αλλιώ μιλούμε για μεγάλη απώλεια εμπιστοσύνη εάν δεν λειτουργήσει το σύστημα ETS, το Emission Trading System. Ευχαριστώ και Έντελμπέκε λοιπόν για την ενημέρωση. Νομίζω ότι θα παραμείνετε εδώ μαζί μας για την συζήτηση που θα διεξαχθεί αργότερα για το 20 ή το 30% και έρχομαι τώρα στο θέμα 3, τα πρακτικά, δηλαδή στις 27 και 28 Οκτωβρίου, επίσης, ε, συγγνώμη, Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις τότε θεωρώ ότι εγκρίνονται. Μετά έρχομαι στα σημεία 5 έως 9, 4 συγγνώμη έως 9, που θέμα είναι η απαλλαγή για το 2009. Έχουμε συγγήτρια ε, που είναι η κυρία Γιούτα Χάουκ και θα μας πει τι στάση πρέπει να τηρήσουμε. Ναι, ευχαριστώ. Ως Επιτροπή Περιβάλλοντος συντάσσουμε γνωμοδότηση και όχι βέβαια την ίδια την απαλλαγή γνωμοδότηση για την Επιτροπή, για λογαριασμό δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού η οποία Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού δύναται να περιλάβει την γνωμοδότησή μας, αλλά τέλος πάντων ίσως χρειαστεί και λίγο σπρόξιμο από πλευράς μας. Το λέω αυτό για να το έχετε υπόψη σας. Εξετάζοντας τώρα τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι θέματα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων. Εξετάζοντας ολόκληρο τον πίνακα θα δούμε ότι στο σύνολο είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά απορρόφησης και σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων, δηλαδή όσα έχει διαθέσει η Κομισιόν με την υπογραφή συμβάσεων και έχει συμφωνήσει δηλαδή με τις χώρες μέλη Συνολικά είναι καλύτερα τα αποτελέσματα το 2009 από ότι το 2008. Όλα αυτά τα ποσοστά αυξήθηκαν. Στον τομέα του περιβάλλοντος κατά, στο, κατά 2% παραπάνω δηλαδή, έφτασαν στο 97,1% Στον τομέα της υγείας σχεδόν φτάνουμε στο 100%. Εάν είχαμε πραγματικά 100% θα έπρεπε να ψάξουμε κάπου το λογιστικό σφάλμα. Και για την ασφάλεια τροφίμων είμαστε στο 98%. ενώ πάντα για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Για τις πιστώσεις πληρωμών, επίσης τα πράγματα πάνε καλά σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την υγεία, σχεδόν στο 100% για το περιβάλλον και μάλιστα 99,92% για την υγεία. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, φτάνουμε μόνο στο 82% απορρόφησης των πιστώσεων πληρωμών εδώ πρέπει να εξετάσουμε βέβαια πού οφείλεται αυτό. Και εάν δούμε ότι στην ασφάλεια τροφίμων συχνά οι υποχρεώσεις βασίζονται στις εκτιμήσεις των χωρών μελών και έτσι αναλαμβάνονται αυτές οι υποχρεώσεις, δηλαδή συμφωνούνται τα ποσά αυτά με τις χώρες μέλη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά οι χώρες μέλη καλούνται να υποβάλουν τους πραγματικούς λογαριασμούς και οι χώρες μέλη κάθε φορά αποδεικνύεται ότι είχαν υψηλά υπερβολικές προσδοκίες. Έτσι τελικά από τις υποχρεώσεις οι πληρωμές καταλήγουν να είναι μόνο στο 82%. Άρα αυτό που πρέπει να ζητηθεί από τις χώρες μέλη είναι να κάνουν ακριβέστερες, ακριβέστερους σχεδιασμούς. Για παράδειγμα για, τον, ε, για τη νόσους των χείρων ή για την γρήπη α1 ή τα 1 και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο ακριβείς υπολογισμούς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δεν ευθύνεται σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες πιστώσεις υποχρεώσεων, αλλά δεν κατέληξαν όλες στο να πληρωθούν. δεν χρειάστηκε να ε, γίνουν όλες αυτές οι πληρωμές. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να μιλήσει κανείς με τις χώρες μέλη. Κάτι που πήγε καλά είναι το πρόγραμμα μας, το πρόγραμμα LIFE. Και εδώ πραγματικά θα πρέπει να επενέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. γιατί, διότι έφτασαν σε ποσοστό απορροφητικότητας 99,9%. Δηλαδή πάλι φτάνουν σχεδόν στο 100%. <clears throat> ίσως να μην θεωρηθεί σπουδαίο αυτό, αλλά θα θυμάστε ότι για το έτος 2009 είχαμε ζητήσει να εγγραφούν 29 εκατομμύρια παραπάνω στο κονδύλι του LIFE από αυτά που είχε ζητήσει στο προσχέδιό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένω, ξαφνικά η Κομισιόν αναγκάστηκε να έχει στη διάθεσή της για να τα διαθέσει 29 εκατομμύρια και κατάφερε να τα βρει. Το 2009 ανελήφθησαν υποχρώσεις για 210 έργα στον τομέα του LIFE για την βιοπικιλότητα ε, περίπου 80, 115 για τη βιοστατηγική και 11 για την επικοινωνία και ενημέρωση. Αυτά είναι λοιπόν σπουδαία νέα και ελπίζουμε το ίδιο υψηλό ποσοστό να φτάσουμε και για το 2010. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την προσπάθεια που, κατέλαβε, που κατέβαλε μάλλον, η ε, Κομισιόν, ε, η πρότασή μου είναι να δοθεί απαλλαγή. Σε ό,τι αφορά τώρα τους οργανισμούς, θα τα πω τώρα κάπως ε, σαρώνοντας όλο τον ορίζοντα, επομένως μιλώ για τον οργανισμό περιβάλλοντος, για τον οργανισμό χημίας, για τον οργανισμό ασφάλειας, την ECDC στο Ελσίνκι και τον Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο. Για όλους αυτούς τους οργανισμούς προτείνω επίσης απαλλαγή, διότι οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, που σημαίνει οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου και οι απαντήσεις των οργανισμών στα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου, Όλα αυτά επιτρέπουν την εξαγωγή του συμπεράσματος ότι δικαιολογείται η πρόταση απαλλαγής των ε, διευθυντικών στελεχών. Τώρα, για όλους τους οργανισμούς, εκτός από την ΕΦΣΑ, ασφάλεια των τροφίμων δηλαδή, θα πρέπει επίσης να λεχθεί ότι τουλάχιστον σε 10 ή και στους 11 οργανισμούς πρέπει να ε, προσέξουν να τηρήσουν την αρχή του ενιάυσιου του προϋπολογισμού, δηλαδή του ετήσιου του χαρακτήρα. <clears throat> το, το, ε, την παρατήρηση κάνει και το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά βέβαια υπήρξαν διάφορες δικαιολογίες ο πλευράς οργανισμών για ποιο λόγο δεν ε, μπόρεσαν να αναθέσουν όλες αυτές τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Το επόμενο στρατηγικό πρόγραμμα θα ψηφιστεί το 2013 για την ΕΚΑ, το, τον οργανισμό ΕΚΑ δηλαδή. Τα προγράμματα που θα προέκυπταν ε, μετά το τέλος της πρώτης περίοδου καταχώρησης ε, πρόκειτο να αρχίσουν. Είχαν γίνει και σχετικές ε, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, αλλά δεν είχαν ακόμα ανατεθεί όλα αυτά τα έργα και επομένως αυτό μπόρεσε να γίνει μόλις στις αρχές του 2010. Για τον οργανισμό ECDC είναι ιδιαίτερα ε, βαρύ το θέμα διότι πρόκειται για θέματα κτηρίων κλπ. Και παραπάνω από 30% του τίτλου 3 αναγκάστηκαν να περάσουν στο επόμενο τους. Τώρα για το τίτλο 2, για τα κτίρια δηλαδή, γνωρίζουμε ότι ο ECDC δεν πρόκειται να ανακαινήσει πλέον ούτε να διαμορφώσει το κτίριο το οποίο κατέχει ήδη, ανταυτού θα μετακομίσει σε άλλο κτίριο, διότι οι συνθήκες για την ανακαίνιση αλλά και η νέα μισθωτική σύμβαση ήταν δυσανάλογα ακριβά. Και έτσι είπε ο διευθυντής του οργανισμού αυτού, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε. Τέρμα εδώ, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ένα νέο κτίριο. Γι' αυτό και δεν δόθηκαν πλέον, δεν διατέθηκαν πλέον κονδύλια για οποιαδήποτε ανακαίνιση. Και για τον οργανισμό του Λονδίνου, ΕΜΕΑ, δεν διατέθηκαν κονδύλια ύψους 38% του τίτλου 2 και έγινε μεταφορά του στο επόμενο έτος διότι υπήρχαν συμβα... είχαν μάλλον λήξει πολιετή συμβάσεις για την παροχή εξοπλισμού ή έτρεχαν ακόμα οι συμβάσει αυτέ, αλλά δεν είχαν ακόμα ε, παραδοθεί όλα τα υλικά αυτά άρα δεν μπορούσαν και να πληρωθούν ώστε χρειάστηκε να γίνει μεταφορά στο έτος 2010. Με λίγα λόγια εν τέλει, όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν λόγο για να αρνηθούμε την χορήγηση απαλλαγής. Όλοι οι οργανισμοί εξετέλεσαν το έργο για το οποίο έχουν ιδρυθεί και μάλιστα γενικά σε καλό επίπεδο. Πρώτος στην τάξη μαθητής είναι η, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και διότι μας έχει πάντοτε τηρήσει ενήμερους με ακριβή στοιχεία και αυτό που θα έπρεπε ίσως να λεχθεί σε όλους τους οργανισμούς είναι η ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας. Και προς την κατεύθυνση του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και προς την κοινή γνώμη. Οι οργανισμοί αποτελούν μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής διοίκησης και μάλιστα και τα τμήματα εκείνα που είναι εγκατεστημένα εκτός Βρυξελών, Λουξεμβούργου, Στρασβούργου. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάπου κάνουν επικοινωνια, επικοινωνιακή πολιτική, είναι λίγο και οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέρη όπου βρίσκονται και επομένως πρέπει εκεί να προσφέρουν περισσότερο και καλύτερο έργο ώστε να γίνονται ορατοί κιόλα και στις χώρε μέλη που βρίσκονται. Έπαινο αξίζει ακόμα στην ΕΦΣΑ, τον, την οποία επένεσε και το ελεγκτικό συνέδριο, τη είπε ότι τα έκανε άψογα με ξεχωριστή εγγραφή στον προπολογισμό για την πρόθεση της έρευνας και για τα επιδόματα που λαμβάνει ούτως ή άλλως από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ξέρω ότι στην Επιτροπή Ελέγχου προπολογισμού, δύο τουλάχιστον οργανισμοί έχουν κληθεί να παρουσιαστούν και ένας από αυτούς είναι μεταξύ των πέντε για τους οποίους είμαστε αρμόδιοι εμείς. Κλήθηκαν οι οργανισμοί αυτοί διότι προφανώς είχε την εντύπωση η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ότι υπήρχαν σε υψηλό βαθμό κάποιες ανομαλίες από πού τώρα έχουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού τις πληροφορίες αυτές. Από τον εσωτερικό οικονομικό έλεγχο της Κομισιόν, το internal audit, το οποίο όμως δεν διαθέτουμε εμείς. Ούτε μάλιστα εγώ που είμαι και η εισηγήτρια για την γνωμοδότηση, ούτε μου επιτρέπεται καν να την δω. Δεν υπάρχει καν αυτό το μικρό δωματιάκι όπου η δυνατότητα δηλαδή να πάει κανείς σε αυτό το μικρό γραφείο που είναι κλειστό και μπορεί να εξετάσει, ε, να διαβάσει κάποιο έγγραφο εμπιστευτικό. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι πάλι εκόντες άκοντες να ακούσουμε τι μας λέει ο εισηγητής τους και εάν μας δώσει τις σωστές πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει από αυτό το internal audit. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να αναλάβουμε μια δική μας πρωτοβουλία στο σύνολό μας ως Επιτροπή και να βγούμε και να πούμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε το έγγραφο αυτό, ε, εάν δεν το λαμβάνουμε, εάν δεν μας διαβιβάζεται. Α, κάτι ξέχασα, αγαπητέ Πρόεδρε. Ε, είδα τον Φλόρενς και το θυμήθηκα. Υπάρχουν βέβαια τα χόμπι του καθενός. Ξανάρχομαι λοιπόν στην ανάγκη πληροφόρησης. Όσα πράγματα είχαν σχέση με μη κρατικού οργανισμούς μπορεί να τα δει κανείς την ιστοσελίδα της ε, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Κομισιόν. Όχι μόνο τα κονδύλια που ε, πήραν, αλλά και το τι ακριβώς κάνουν. Αυτά λοιπόν. Σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες προς τον Καρλ Χάιντς ε, Φλόρενς. Τα σημειώνουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε Γιούτα Χάουγκ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 11 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι και θα πρέπει τον Μάρτιο να ψηφίσουμε προς έγκριση. Έχουμε όμως ακόμη μία παρέμβαση. Τόμας Ούλμα, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πω ότι τη χορήγηση απαλλαγή για τι υπηρεσίε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επιμέρου τμήμα 3 θα την υπερψηφίσουμε. Σίγουρα οι υπηρεσίε ε, ζουν στον δικό τους μικρό κοσμό, μακριά από τις Βρυξέλλες και έτσι έχουν είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς μια πλήρη επισκόπηση και να ελέγξει τα πάντα. Σημαντικό είναι η internal audit, δηλαδή η εσωτερική έλεγχη, να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να γνωρίζει κανείς, είναι κάτι αυτονόητο όταν βλέπει κανείς πόσο με διάφανο τρόπο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να αναμένουμε το ίδιο να ισχύει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ 104 νέες ε, θέσεις που δημιουργούνται για την ΕΦΣΑ. Και όλα αυτά λειτουργούν σχετικά καλά για την ECD. E Είναι κατανοητό ότι έχουμε εδώ το πρόβλημα του ότι το ίμιση του ποσού δεν δαπανήθηκε εμπρόθεσμα και έχουμε ένα υπόλοιπο κάποιων εκατομμυρίων που απομένει ακόμα. Δεν αναφέρονται τώρα όλα τούτα, αλλά όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν ε, ε, βρεθεί καλά, καλώς. Τώρα έχω δει εδώ και ένα σφάλμα όσον αφορά την ε, τεκμηρίωση που λείπει. Έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ που είναι εδώ. Για το τρίτο τώρα τμήμα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να πούμε ότι το ποσοστό εκτέλεσης με 97,12% είναι πολύ ικανοποιητικά αυτά τα ποσοστά και θέλω θετικά να αναφέρω αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Ποιος θα ήθελε ακόμη να παρέμβει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν υπάρχει κάποιος. Λοιπόν, όπως είπαμε, 11 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Και θα μπορεί κανείς ε, και τις ε, τροπολογίες για την έκθεση Utah Hawk να τις καταθέσουμε. Έτσι ευχαριστούμε Utah για αυτή τη δουλειά που κάνεις ε, για λογαριασμό της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Είμαστε ευγνώμονες. Κάποιος πρέπει να, έχει, να εξοικειώνεται και να μπορεί να ελέγξει και να δει τι γίνεται με αυτά τα στοιχεία, θετικά ή αρνητικά. Αυτά είναι τα, στοιχεία 4, τα σημεία 4 έως 9. Φτάσαμε στο σημείο 10 λοιπόν. Έκθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διάσκεψη για τις κλιματικές, κλιματολογικές αλλαγές στο Κανκούν. Η έκθεση είναι στη διάθεσή σας επί τραπέζης, την έχετε διαβάσει όλοι και στο Στρασβούργο εξάλλου. Μετά το Κανκούν είχαμε συζήτηση που διεξήχθη σχετικά. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τη γραμματεία μας, τον Γιώργο Αμανατίδη και τους συναδέφους που στην προπαρασκευή και διοργάνωση μιας τέτοιας εβδομάδας συμμετείχαν για την διάσκεψη του ΟΗΕ. Όλα αυτά στην Κοπεχάγη λειτουργήσαν πολύ καλά. Είχαμε ένα ευρύτατο πρόγραμμα με κοινέ συναντήσεις ε, με συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια και σε σχέση με το Μεξικό, Νότια Αφρική, Βραζιλία, με οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και την Παγκόσμια Τράπεζα και φυσικά με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με ΜΚΟ. Θα έλεγα ότι η ενημέρωση από την Επιτροπή, οι ενημερωτικές συναντήσεις από την Επιτροπή και το Συμβούλιο ήταν καλές. Και στο τέλος είχαμε κάποια προβλήματα χρόνου, χρονικά προβλήματα, πίεζε ο χρόνος. Πρέπει κανείς να δεχθεί αυτή την κατάσταση. Οι τελικές διαπραγματεύσεις ε, ε, είχαν τέτοια μορφή που πίεζαν πολύ ήταν καλό αυτό και το βρήκαμε θετικό διότι στη διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών κάποιοι, κάποιες επιτροπές ε, άσκησαν ε, υπέβαλαν παράπονα για την συμμετοχή και την ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου σε διεθνείς συναντήσεις. Ούτε για το Κανκούν ούτε για την Αγκόγια θα μπορούσαν να συμμεριστώ τέτοιες επικρίσεις. Ήταν καλές αυτές οι εκδηλώσεις. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε όλοι. Τίθεται το ερώτημα ποια συνέχεια θα δοθεί ώστε να έχουμε το Δεκέμβριο τη συνέχεια που θα ακολουθήσει. Θα έχουμε και το απόγευμα αυτή τη συζήτηση για την έκθεση αν θα έχουμε σχετικά 20-30% μείωση των εκπομπών ρήπων. Τα ουσιοδέστερα προβλήματα έρχονται ακόμα, βρίσκονται μπροστά μας. Μια δεσμευτική νομική βάση για μια τέτοια ε, σύμβαση, για μια τέτοια συμφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος και για το Κιώτο μετά το Κιώτο και όσα συνδέονται ως θέματα και ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο μείωσης ε, των εκπομπών ρήπων. Αυτά που έχουμε επιτραπέζεις δεν επαρκούν ως προτάσεις. Το γνωρίζουμε αυτό. Μεταξύ τριών και 3,5 βαθμών Κελσίου κινούμαστε και στο Κανκούν είχαμε ένα μείζωνα αποτέλεσμα ως συμπέρασμα ότι συμφώνησε η διεθνής κοινότητα να επιτρέψει μόνο 2 βαθμούς Κελσίου στην υπερθέρμανση, στην θέρμανση του πλανήτη. Είμαστε πολλές αντιπροσωπείες και μετά από έντονες διαπραγματεύσεις υπήρχαν και, υπήρξαν και άλλοι συνάδελφοι που ε, συμμετείχαν. Στην Κοπενχάγη ήταν 72, ήταν λιγότεροι δηλαδή στο Μεξι... από ό,τι στο Μεξικό. Και το συνολικό αυτό πλαίσιο μπόρεσε να ταιριάξει πολύ καλά σε σχέση με τις συναντήσεις ε, που είχαμε και πρέπει να δούμε πώς θα προπαρασκευάσουμε την επόμενη κορυφή, σύνοδο κορυφής για αυτό το θέμα. Λοιπόν, εσείς κύριε Γιάνγκιασεν, παρακαλώ. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα και εγώ θερμά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της γραμματείας μας ε, που είχαν συμμετάσχει και συμμετείχαν στο Κανκούν. Το πρόγραμμα ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Πιστεύω ότι βρήκαμε μια καλή ε, γραμμή. Αφενός εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα πολύ ενδιαφέροντες ε, ενδιαφέρουσες προσωπικότητες να συναντήσουμε. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία που προσφέρεται σε σχέση με ΜΚΟ, οργανώσεις ε, του οργανισμού του ΟΗΕ και πολιτικούς. Είχαμε λοιπόν πολύ καλές τέτοιες συναντήσεις. Αυτή είναι η μία πλευρά. Το άλλο όμω είναι το ότι και εμείς ως Κοινοβούλιο μπορέσαμε να ασκήσουμε και την επιρροή μας. Διότι σε σχέση με την δική μας αντιπροσωπεία συναντήσαμε και εθνικούς βουλευτές που στο πακέτο για τα μέτρα για το κλίμα εξειδικευμένο νομοθετικό έργο είχαν εκπονήσει και είχαν προτείνει. Μπορούμε πραγματικά να επενέσουμε αυτή την εκδήλωση και αυτή, αυτές τις εκδηλώσεις. Ε, μπορούμε υποδειγματικά να συνεργαστούμε, να εργαστούμε και να ε, συμμετάσχουμε και εμείς ε, λέγοντας στους άλλους πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα σε σχέση με μας. Μαθαίνουμε και εμείς από τους άλλους. Πρέπει λοιπόν να επενέσουμε και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες και τις ενημερωτικές συνεδριάσεις παρόν σε αρκετέ συναντήσει ε, ΚΟΠ και ποτέ δεν είχαν λειτουργήσει τα πράγματα τόσο καλά όσο αυτή τη φορά. Η Επίτροπος Εντεγκόντ έδωσε πολύ καλές πληροφορίες, ουσιώδεις ε, βασικές πληροφορίες και αυτό ήταν θετικό. Για ένα πράγμα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες εμείς ακόμα από πλευράς μας. Το θεωρώ πραγματικά ότι δεν επαρκεί, λέγω, ότι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στις ομάδες συντονισμού του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μη συμμετέχει. Έχουμε καθεστώς παρατηρητού. Σωστό αυτό, αληθεύει. Όμως το καθεστώς παρατηρητού θα έπρεπε να σημαίνει ότι τουλάχιστον ο πρόεδρος της δικής μας αντιπροσωπείας, όχι το σύνολο της αντιπροσωπείας, φυσικά αλλά ο πρόεδρος μας πρέπει να συμμετέχει και να είναι παρόν όταν θα συζητούνται θέματα της ε, πολιτικής για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Και πολλοί συμφωνούν και λένε ότι αυτό ήταν ένα μέρος Τη συμφωνίας πλαισίου. Και γι' αυτό ήταν αυτός ένας λόγος που υποστηρίξαμε τον Παρόζο και είπαμε ότι εντάξει, ωραία, εμείς πρέπει να εγκρίνουμε διεθνείς συμφωνίες, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα συμμετέχουμε στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και έγκρισης αυτών των συμφωνιών. Και εδώ δεν βλέπω το πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εκπροσωπείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια και ούτως ή άλλως ως παρατηρητές είμαστε παρόντες από το Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά τον μελλοντικό προγραμματισμό και σχεδιασμό για την Νότια Αφρική, θα έλεγα ότι προσωπική μου άποψη είναι ότι εμείς όχι μόνο θα πρέπει επί της ουσίας ε, και επί του περιεχομένου να συζητούμε και αυτό το κάνουμε επί πολύ χρονικό διάστημα και γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιθυμίες και ε, οι στόχοι του Ευρωκοινοβουλίου. Κάτι τώρα θα πρέπει περισσότερο, περισσότερο να επικεντρωθούμε στα εσωτερικά θέματα ως Κοινοβούλιο έναντι των άλλων θεσμικών οργάνων. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος Χέντεγκορ ε, όντας ε, ανοιχτή και δείχνοντας πνεύμα συνεργασίας πρέπει να, είναι, να δειχθεί συνεργασία και γι' αυτό το σημείο θα ήθελα όχι μόνο επί της ουσίας να επικεντρωθώ για αυτό το θέμα, μια και έχουν συζητηθεί και αυτά στο Στρασβούργο, αλλά για άλλη μια φορά θα ήθελα να συνεχίσω στην παρέμβαση του ε, Προέδρου στα όσα είπε. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η δουλειά και θα ήθελα να μπορέσει κάποιος να μου εξηγήσει πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν ακόμα καλύτερα. Ήταν λοιπόν πολύ καλά τα πράγματα και ήταν ευχάριστο το κλίμα, θετικό το κλίμα και είδαμε ότι υπήρχε κίνηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, αν τα καταφέρετε με τους συνεργάτες σας να συνεχίσετε αυτή τη θετική πορεία με τη γραμματεία, μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας εκφράσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Χαίρεται κανείς πάντα για επένους. Θα το διαβιβάσω αυτό και διαβιβάζω αυτούς τους επένους τους συνεργάτες μας που διοργάνωσαν αυτά τα πράγματα με αυτό το θετικό πνεύμα. Ο Κρήτον παρακαλώ, Κρήτον Ασένης παρακαλώ. Thank you very much, Mr. President. Uh... It was indeed a very successful. Πράγματι ήταν μια πολύ επιτυχής αντιπροσωπεία. Και ήταν επίσης μια ιδιαίτερος επιτυχής συνάντηση σε σχέση με αυτά τα οποία μπορούσαμε να φοβόμασταν. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω αφορά τις αντιπροσωπείες. Την επόμενη φορά θα πρέπει να διευρυνθούν όσο περισσότερο γίνεται η διάρκεια τους μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης. Και για την Αγκόγια και για το Κανκούν, τη νύχτα που γινόντουσαν οι βασικές διαπραγματεύσεις, πολύ λίγοι από εμά μπόρεσαν να μείνουν μέχρι το τέλος. Θα πρέπει να παραταθούν λοιπόν οι αντιπροσωπείες μέχρι και το τέλος των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να πω επίσης κάτι άλλο. Κάτι το οποίο δεν συζητιέται ιδιαίτερα. Τη νύχτα των διαπραγματεύσεων ένα πολύ δύσκολο θέμα τέθηκε προς συζήτηση. Η Βολιβία έλεγε όχι στο τελευταίο, στο τελευταίο λεπτό και η απόφαση ελήφθη χωρίς τη Βολοβία παραβιάζοντας τους κανόνες λήψης των αποφάσεων, που πρέπει να είναι ομόφωνες εννοεί ο κ. Αρσένης. Αυτός ο κανόνας ε, κατερρίφθη στο Κανκούν. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο μέλλον. Συμφωνώ πάντως ότι έχουμε πλέον μια απόφαση και οι διαπραγματεύσεις θα επηρεαστούν από αυτήν στο μέλλον. Thank you, σε ευχαριστώ Κρήτον. Θα έλεγα η Μεξικανική Προεδρία ερμήνευε τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών και δεν τους παραβίαζε. Εγώ πιστεύω ότι πολύ καλά πήγαιναν τα πράγματα και ήταν σωστό η συμφωνία του Κανκούν με αυτόν τον τρόπο να τεθεί και ήταν ερμηνεία του TST συνένεση σχετικά. Και επενώ λοιπόν για αυτό το επίτευγμα και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα πορεία στο μέλλον της διαπραγματεύσεις ε, των Ηνωμένων Εθνών και τη διαμόρφωση διαδικασιών και διεργασιών συνένεσης. Λοιπόν, εντάξει. Μαρίτα Ουλσκοκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Eh, eh, ett möte som eh, gjorde skillnad εγώ, η συνάντηση αυτή επέτρεψε πράγματι να κάνουμε θετικά βήματα. Στην αρχή η αίσθηση ήταν ότι βαδίζαμε προς το αδιέξοδο, αλλά δεν υπήρξε καταστροφή, δεν υπήρξε αδιέξοδο. Καταφέραμε να κερδίσουμε χρόνο και πλέον σε αυτή τη φάση έχει σημασία να διαπιστώσουμε ότι έχουμε κάποια μέσα για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση και αυτό θα συμβεί στη συνάντηση του Ντέρμπαν. Συναντηθήκαμε και με την αντιπροσωπεία για την Νότιο Αφρική και η αντιπροσωπεία αυτή νομίζω ότι έχει αρκετές ε, προσδοκίες σχετικά με τη συμμετοχή και τον ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να παίξουμε ένα σημαντικότατο ρόλο στον Τέρμπαν. Έχουμε τη δυνατότητα εφόσον θέλουμε τον Τέρμπαν να αποτελέσει τη συνέχεια των προσπαθειών μας μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα κερδίσαμε απλά χρόνο Τώρα όμως ε, έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις στη διάθεσή μας και νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας στον Τέρμπαν. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σε δύο σημεία θα ήθελα να πω κάτι. Αφενός στο θέμα, στο θέμα της διοργανικής συμφωνίας πλαισίου. Ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις και το θέμα της συμμετοχής του Ευρωκοινοβουλίου, εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου σε διεθνείς τέτοιες διασκέψεις ήταν πιθανότατα το πιο επίμαχο θέμα από όλα. Οι απόψεις σχετικά ήταν πραγματικά ασυμβίβαστες μεταξύ τους. Παρόμοια όμως πρέπει να πω ότι η αναγκαιότητα εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις συνεδριάσεις αυτές να συμμετέχουν εδώ σε μας στο σύνολο της Ευρωβουλής δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως εγώ τα βλέπω τα πράγματα εντάξει όπου και εκεί πάντα γίνεται, θα γινότα, γίνεται η διαφοροποίηση ποιου είδους αυτές οι διασκέψεις είναι και η επιθυμία, πρέπει να πούμε ειλικρινά υφίστατο, να διαφοροποιούνται μεταξύ διαπραγματεύσεων που διεξάγει ως υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου θέλουμε και ενδεχόμενα το τελικό αποτέλεσμα να υφίσταται επικρίσεις και της μη συμμετοχής του Ευρωκοινοβουλίου. Πάντα τονίζουμε και λέμε ότι πρόκειται για καθεστώς παρατηρητού και ότι οι διαπραγματεύσει ε, με αυτόν τον τρόπο από πρώτο χέρι μπορούν να κριθούν από εμάς. Αλλά σε διατυπώσεις που βρίσκονται στο τελικό κείμενο υπάρχει κάποιο περιθώριο εκτίμησης για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησης επιρροή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σίγουρα σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφοροποιούνται τα πράγματα για την προθυμία να γίνονται αυτά με τον έναν ή άλλο τρόπο για τον τομέα του εμπορίου ή τον τομέα του περιβάλλοντος. Αλλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ίσως κάποιοι θα ήταν πρόθυμοι εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, όχι μόνο αναγκαία τον πρόεδρο ή την πρόεδρο σε σχέση με την αντιπροσωπεία. Μια αντιπροσωπεία να μπορούσε να συμμετέχει με δύο ή τρία άτομα από το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετέχει μια τέτοια αντιπροσωπεία. Ήταν όμως ε, ισχυρή αντίσταση, ε, η αντίθεση του Κοινοβουλίου. Και ήταν απόλυτα σαφές ότι οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, με συγχωρείτε, του Συμβουλίου που ήταν αντίθετοι, εμένουν και επιμένουν να υπάρχει μια ξεχωριστή, ένα ξεχωριστό πλαίσιο όπου δεν θα συμμετέχει το Ευρωκοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις αλλά θα παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και τα αποτελέσματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν το δει κανεί, αυτό είναι το τμήμα, αυτό το οποίο είναι το πιο αδύναμο από όλους τους κρίκους. Θα ήθελα μια σύντομη παρατήρηση επί της ουσίας να κάνω για το ίδιο το θέμα. Διαπιστώνω επανειλημμένα πάντα ότι σε διεθνείς συνδιασκέψεις σε σχέση με τη συμμετοχή που λόγω αρχής ε, δεν το κάνω. Τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε να διαμορφώνονται από κάποιους ε, που συμμετέχουν ή διαβάζοντας από τον τύπο, από τα αποτελέσματα μου φαίνονται κάπως διαφορετικά από εκείνα τα αποτελέσματα τα οποία μας ανακοινώνει η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι η εφορία να συμμετέχει κανείς σε αυτό το πλαίσιο και κάπως να μπορεί κάτι να πετύχει, καμιά φορά μας κάνει να ξεχνάμε την ίδια την πραγματικότητα και να μην την λαμβάνουμε υπόψη. Και εν κατακλείδη αυτού του είδους οι εκθέσεις όπως ε, και στο ε, στο Προεδρείο έχουν αναφερθεί τα σχετικά. Το βρίσκω αυτονόητο. Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος που είναι υπεύθυνα και είναι υπέρ μιας πολιτικής για τα κλιματικά θέματα να προσπαθούν να, να ζουν με ουδέτερο τρόπο, ας το πω έτσι όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων, στα ταξίδια και αποστολές που συμμετέχουν. Εγώ το κάνω και είναι αυτονόητο αυτό. Ο Νταν Γιώργενσεν και άλλοι και εκείνοι το κάνουν. Καλύτερο όμως θα ήταν και πιο ωραίο αν υπήρχε μια άλλη δυνατότητα από το να πηγαίνουμε σε αυτά τα ταξίδια δηλαδή να παρακαλάμε το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να εγκρίνει μια αποστολή σε μια διάσκεψη για το κλίμα και να γίνεται αυτό εις βάρος του Κοινοβουλίου. Το βρίσκω πραγματικά αξιοπερίεργο να ζητά κανείς να κάνει κάτι και το Κοινοβούλιο να μην συμμετέχει βλέπουμε συνολικά ποιες είναι οι δυνατότητες να υπάρχει ουδετερότητα όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα ταξίδια και τις αποστολές για τους ευρωβουλευτές και άλλους. Πρέπει ειλικρινά να πω ως πολιετές μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είδα το αίτημα και ντράπηκα. Είναι η δεύτερη φορά που ντράπηκα με κάτι τέτοιο και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Καλύτερο θα ήταν πρωτού περάσει στο Προεδρείο αυτό το αίτημα να συζητούσαμε με τους συντονιστές αν θα ήταν αναγκαίο ή όχι να κατατεθεί έτσι. Ευχαριστώ. Ροσμπαχ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσέξτε. Θα ήθελα να αποφύγω να επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα που προαναφέρθηκαν. Θέλω όμως να ευχαριστήσω θερμά τη Γραμματεία για το ότι με αυτόν τον καλό τρόπο ε, διοργάνωσε τα πράγματα. Ξέρω δεν είναι παρούσα η κυρία Χέντεγκάρντ αλλά μας ενημέρωσε πάρα πολύ θετικά και χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στο τέλος υπήρξε και κάποιο έγγραφο, ένα κείμενο το οποίο ε, ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Θα προτιμούσα όμως φυσικά αν αυτό το έγγραφο είχε και περισσότερο πρακτικά πράγματα τα οποία θα εμπεριείχε ή θα ήταν περισσότερο σαφές ας το πω έτσι. Θα το προτιμούσα αν γινόταν αυτό. Και για το 10 στην Αγκόγια και για το πανεπιστήμιο που δεν αναφέρεται στο έγγραφο και αυτή είναι η βάση για τη συζήτησή μας συνολικά για τα κλιματικά, κλιματολογικά θέματα. Η βιοπικιλότητα, με συγχωρείτε, η βιοπικιλότητα πρέπει να είναι με σαφήνεια ένα θέμα το οποίο θα εμπεριέχεται. Και το, η, σχέση σε, ε, η συμμετοχή των ηθαγενών λαών. Αφενός θέλουμε να προστατέψουμε το περιβάλλον με κάθε τρόπο σε όλα τα επίπεδα. Το νερό, τα ύδατα, τα δάση, από την άλλη όμως πλευρά πρέπει και τρόφιμα να παράγονται για 6,5 δισεκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη. Και αυτός ο αριθμός των κατοίκων του πλανήτη αυξάνεται και μάλιστα με, ισχυρή, με ισχυρό ρυθμό αύξησης. Θέλω να δω πώς θα τα καταφέρουμε. Δύο παρεμβάσεις λέει ο πρόεδρος και μετά κλείνει ο κατάλογος αγορητών. Και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ματία Φροντίνο, επόμενος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία διάσκεψη αφενός και τώρα είχαμε και συνεχώς και διαρκώς ε, ε, στον χώρο επισκεπτών ε, χώρο και θέση και είχαμε αυτή την συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και εκεί πρέπει να επιμείνουμε και να εμείνουμε ως Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στις επόμενες διασκέψεις να είναι σαφές ότι ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου θα βρίσκονται άμεσα και θα είναι παρόντες στους χώρους όπου γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Πάντα το Κοινοβούλιο πρέπει να πούμε ότι δεν κατανοεί γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε και να ασκήσουμε την επιρροή μας ε, όταν πρόκειται για τέτοιες αποφάσεις το Κοινοβούλιο να βρίσκεται πρώτο-πρώτο μπροστά-μπροστά στις γραμμές, στις σειρές ε, των παρόντων. Διότι διαφορετικά σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις δεν θα είχαν νόημα. Σίγουρα είναι αξιόλογο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να μπορεί κανείς να συμμετέχει, επιστρέφει με πολλά βιώματα και πολλές ε, θετικές εντυπώσεις, αλλά παρακαλώ να ασκήσουμε την επιρροή μας, να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να συντάξουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας στο γύρο των ε, Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ε, να δούμε τι γίνεται σε άλλες ε, διεθνείς διασκέψεις ε. αν έτσι μπορεί να δοθεί συνέχεια. Είναι σαφές ότι με τη Λισαβόνα, συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε μια νέα περίοδο, μια νέα εποχή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος ε, ως συμμετέχον, ως εμπλεκόμενο όργανο με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και όσον αφορά αυτά τα οποία ανέφερε η συνάδελφος Ροτ Μπέρεντ, είναι αυτονόητο για έναν πολιτικό που ασκεί την επιρροή του για θέματα περιβάλλοντος με αυτόν τον τρόπο να τοποθετείται διότι εδώ πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα, να δίνουμε πάντα το καλό παράδειγμα και να προβληματίζει το καθένας να δει πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Ευχαριστώ. Συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε ε, τέτοιες διεθνείς διασκέψεις είναι μόνιμο θέμα για τη διάσκεψη των Προέδρων μπορώ να πω Χρειάζεται μια σωστή συμφωνία, ένα σωστό πλαίσιο και αυτό θα μπορεί και για τις άλλες επόμενες ε, συνδιασκέψεις να λειτουργήσει. Προϋπόθεση να υπάρχει μια τέτοια προοπτική για μια τέτοια συμφωνία και να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο και να συμμετέχει με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ο επόμενος αγορητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Dagmar Rothberend για την πρωτοβουλία της, ιδιαίτερα για τον ρόλο των Ευρωβουλευτών και του Κοινοβουλίου σε τέτοιου είδους διεθνείς διασκέψεις. Ο ίδιος ως νομικός γνωρίζω τους κανόνες και τους κανονισμούς σε σχέση με το πώς λειτουργούν αλλά τα γρανάζια, αλλά πρέπει να έχουμε μια δυναμική, ας το πω έτσι, στη συμμετοχή μας και να λάβουμε υπόψη ότι ως Ευρωβουλευτές έχουμε ένα ιδιαίτερο ρόλο στην διαμόρφωση και αποκριστάλλωση απόψεων και για το ρόλο μας ως παρατηρητών είναι σαφές ότι έχουμε αιτήματα και διεκδικούμε συγκεκριμένα θέματα και θα είναι θετικό την, να έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο απέναντί μας θα πρέπει με δυναμικό ενεργό τρόπο να συμμετέχουμε και για την εφορία και το, την πραγματικότητα για το σχόλιο που έγινε έχετε δίκιο σε αυτό αλλά βλέποντας τα μέσα ενημέρωσης ε, και τα δημοσιεύματα πιστεύω ότι εμείς ε, ως υπεύθυνοι πολιτικοί για το περιβάλλον είναι σημαντικό να κινούμαστε και να βασιζόμαστε στα θεμέλια του δικαίου διότι όταν πλησιάζουμε ή προσεγγίζουμε μια συμφωνία ή ένα τέτοιο πλαίσιο, βλέποντας ε, τις, ε, την νομική πραγματικότητα και τα, την, ας το πω έτσι, τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη πραγματικότητα από νομικής πλευράς καταδεικνύεται σαφώς ε, ποια είναι τα όρια και πού βρίσκονται τα όρια σε σχέση με την δυνατότητα να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Και για να έχουμε αυτή την προσέγγιση της πραγματικότητας με ρεαλιστικό πνεύμα είναι σημαντικό να είμαστε σύνετοι ε, και να τηρούμε συγκεκριμένες αρχές, ε, νομικά πλαίσια και να διαφοροποιούμε σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έγιναν για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, θα παρακαλούσα με την ηθικολογία αυτή, η ηθική αυτή διαπαιδαγώγηση να είμαστε πιο ε, σύνετοι και πιο περιορισμένοι. Εγώ θα ήθελα σε σχέση με τα όσα προαναφέρθηκαν να πω ότι στην Αυστρία τέτοιου είδους ε, ηθικά σχόλια ε, πολλές φορές γίνονται και δεν θα ήθελα να γίνονται αυτά δεκτά θεωρώ ότι όταν έχουμε συναδέλφους που τηρούν τους κανόνες, αυτοί δεν είναι ε, λιγότερο καλοί από άλλους. Αυτό λοιπόν ισχύει για όλους, όχι μόνο για μας τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, για κάποιους που τηρούν κάποια πράγματα ή όχι. Είτε είναι δική μας είτε όχι. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι, ολοκληρώσαμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα και πρέπει δύο πράγματα εδώ να παρατηρήσω. Αφενός ο Κρήτον Αρσένης έχει δίκιο ότι είναι πολύ αρνητικό όταν και αν το κοινοβούλιο, ιδιαίτερα τότε, όταν η αντιπροσωπεία του, ας το πω έτσι, έρχεται η ώρα, τα πράγματα και γίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και έχουμε ε, τέτοιες διασκέψεις, στο επίσημο πρόγραμμα να λέγεται τέλος της, ε, της ε, συνεδρίασης ε, αυτό το απόγευμα ξέρουμε ότι στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών ακριβώς το βράδυ η νυχτερινή συνεδρίαση και προς το Σάββατο ήταν η πιο φλέβουσα. Αλλά επίσημα είχε ολοκληρωθεί η αποστολή μας και έτσι δεν υπήρχε τέτοιου είδους, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών παρουσία. Δεν θα είναι δυνατό γραφειοκρατικά να επιτελούμε το έργο μας στη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις και να γυρνάμε μετά να επιστρέφουμε πρόωρα. Έχει μετά ο Γιώργος δίκιο ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει ιδιαίτερο ρόλο και σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει σε εκείνα τα λίγα όργανα που έχει και νομοθετικό έργο που επιτελεί και σε σχέση με τα άλλα κοινοβούλια στην Ιαπωνία, στο Μεξικό, τη Βραζιλία, το είδαμε. Πιο ενδιαφέρον υπάρχει για το πακέτο μέτρων που υιοθετείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το ψήφισμα για το Κανκούν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πολύ θετικό τρόπο σημειώθηκε αυτό το οποίο το Νοέμβριο στην Ολομέλεια είχαμε αποφασίσει για αυτή τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά σε σχέση με αυτή τη σύντομη συζήτηση για αυτή τη ε, διάσκεψη του Δεκεμβρίου. Και τώρα στρέφουμε το βλέμμα στο μέλλον τι, σε σχέση με το τι θα κάνει η κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Φτάσαμε στο σημείο 11, ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων. Να κινηθούμε, να μετακινηθούμε πέρα από το 20% στη μείωση των εκπομπών ρήπων, αξιολογώντας και εκτιμώντας το θέμα διαρροής άνθρακα. Αυτό είναι το θέμα που με την Επιτροπή Βιομηχανίας, την Ήτρε, μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συντάσσεται και ο συντάκτη έγκαιρα είναι παρόν. Παρακαλώ κύριε συντάκτη να λάβετε τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη συζήτηση την οποία κάνουμε γύρω από το θέμα αυτό για το αν θα πρέπει η Ευρώπη να περάσει μονομερό στο 30%. Καιρό είναι πάντω, εμεί σαν κοινοβούλιο να ξεκινήσουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο θέμα. Η Επιτροπή Ήτρε είναι έτσι και αλλιώ αρμόδια επί της ουσία. Έχουμε μια στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ήτρε για κάποια από τα θέματα γιατί έχουν την κύρια αρμοδιότητα σε τομείς όπως η βιομηχανία και η ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι με πνεύμα συνεργασίας θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια καλή έκθεση με την εισηγήτρια επί της ουσίας την κυρία Τζόρνταν. Νομίζω λοιπόν ότι έχει σημασία η στενή συνεργασία μεταξύ μας. Αυτό είναι προς το συμφέρον του συνόλου του Κοινοβουλίου να καταλήξουμε σε μια ισχυρή επιτέλους θέση. Ο χρονισμός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πριν από τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει την άποψή του ένα χρόνο μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο, που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2010. Ένας άλλος λόγος που, επηρεάζει, που επηρεάζεται από το χρονισμό όπως λέγαμε είναι ότι το να πάμε στο 30% είναι κάτι που θα επηρεάσει ε, τα κράτη-μέλη με διαφορετικό τρόπο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της τον μήνα Ιούνιο θα κάνει προτάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν ε, ιδιαίτερα τη συζήτηση. Τώρα περνάω στο θέμα του περιεχομένου. Στον φάκελό σας βλέπετε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο βρίσκεται υπό διατύπωση. Επαναλαμβάνω, είναι έγγραφο εργασίας. Απλά έχω συγκεντρώσει πάρα πολλά επιχειρήματα. Δεν είναι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας, είναι ένα πρώτο κείμενο στα πλαίσια του οποίου συγκεντρώνω όλα τα επιχειρήματα, τις μελέτες, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μία βάση συζήτησης. Είναι λοιπόν μία συγκεκριμένη άποψη και όχι μία επίσημη άποψη του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το έγγραφο εργασίας ακολουθώ την διατύπωση και τη διάρθρωση, αν θέλετε, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. αυτό το κείμενο εργασίας νομίζω μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα εγώ τουλάχιστον να διαμορφώσω την μορφή της έκθεσης τελικά, δηλαδή την πορεία προς το 250, την αποτελεσματικότητα του ETS, το κόστος του μείον 30% και το θέμα της συζήτησης για την απώλεια τη διαρροή άνθρακα να υπογραμμίσω ότι από πλευρά τη ΣΥΤΡΕ θα ασχοληθούν με κάποια από τα θέματα αυτά, όπως οι ανανεώσιμες πηγές, οι βιομηχανικές πολιτικές και θα προσπαθήσουν λοιπόν να προετοιμάσουν την τελική τους έκθεση σχετικά γρήγορα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε σωστά με την κυρία Τζόρνταν. και εγώ θα μεταφέρω το αρχικό αυτό κείμενο στην τελική έκθεση την οποία θα προετοιμάσω επί τη βάση όλων των επιχειρημάτων τα οποία θα προέλθουν και από τη σημερινή συνάντηση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν υπάρξει απόψεις στο παρελθόν, έχουμε συμφωνήσει στο ψήφισμα για το Κανκούν. Είναι σαφές λοιπόν ότι η βάση της έκθεσής μου θα είναι το ψήφισμα το λεγόμενο Κανκούν. Για τα επιχειρήματα. Γιατί τουλάχιστον στην έκθεσή μου θα πω ότι το να περάσουμε στο μείον 30% είναι κάτι το ιδιαίτερα λογικό. Αυτό τεκμηριώνεται από την μακροπρόθεσμη πορεία μας μέχρι το 2050 όπου έχουμε περάσει, ε, έχουμε δεχθεί να φτάσουμε στο μείον 80%. Οπότε είναι πολύ λογικό το 2020 να είμαστε μείον στο 20%. Είναι λοιπόν μια σταδιακή θα έλεγα λογική η οποία θα μας οδηγήσει στην φάση ανάμεσα 25 και 40%. Και γι' αυτό ακριβώς αν συμφωνήσουμε για το 30% ε, είναι κάτι το λογικό, ενώ άλλες προτάσεις ε, δεν είναι. Τώρα, έχουν υπάρξει αλλαγές ε, βέβαια και στις αποφάσεις τις οποίες είχαμε πάρει στο παρελθόν σχετικά με το να πάμε στο 20% μείον και μετά να πάμε στο 30% μείον εφόσον υπάρξει διεθνή συμφωνία. Στα πλαίσια των αποτελεσμάτων του Κανκούν, οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου έχουν δώσει υποσχέθη στα πλαίσια της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να συζητήσουμε τα διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας αν θέλετε, αλλά μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι μεγάλες οικονομίες έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους ήδη από το 2008. Έχει σημασία να προσπαθήσουμε να δούμε και πέραν του Κανκούν, να δούμε σαν παράδειγμα τι προγραμματίσει η Κίνα τον Μάρτιο θα παρουσιάσουν το πενταετές οικονομικό του σχέδιο γιατί πάντα με το σύστημά τους αναφέρονται σε πενταετής κύκλους προγραμματικούς. Κάποιοι είναι υπέρ του συστήματος αυτού, κάποιοι όχι. Εγώ δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα μας προτείνουν στα πλαίσια του πενταετούς ε, σχεδιασμού και νομίζω ότι το πράσινο θα χαρακτηρίζει την οικονομική τους ε, δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο ε, νομίζω έχει νόημα για τους ίδιους, για την οικονομία τους, για το ίδιο τους το έδαφος και το περιβάλλον τους. Λοιπόν, η Κίνα εξελίσσεται αλλά και προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια άλλα θέματα που αφορούν την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. Αν δούμε τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, για μια ακόμη φορά βλέπει κανείς ότι η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες πλήρωσε 70 δις περισσότερα για εισαγωγές πετρελαίου λόγω της αύξησης των τιμών. 70 δις. Γι' αυτό λοιπόν το να γίνουμε λιγότερο εξαρτημένοι από ρηκτά καύσιμα όπως και άνθρακα βέβαια ενώ όχι μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για το ETS, το σχήμα των ανταλλαγών. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του ETS. Να πούμε ότι και εδώ έχουν αλλάξει πολλά από το 2008, σαν παραδείγμα στο τέλος της φάσης 2 θα έχουμε ένα πλεόνασμα γύρω στα 800 εκατομμύρια τόνων διοξίδιου του άνθρακα και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγει ότι ε, το 30% μπορούμε να το πετύχουμε με τα μισά τουλάχιστον πλεονάσματα που μπορούμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν αλλάξει πολλά από το 2008. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο πώς θα πετύχουμε το στόχο του μείον 30% στον τομέα εκτός ETS. Κτηριακή αποτελεσματικότητα στον τομέα της ενέργειας. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θα έλεγα κάνει όλες τις προσπάθειες τις οποίες μπορεί στον τομέα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι αν πετύχουμε το στόχο του 20% ήδη θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Βέβαια στο εσωτερικό του ETS θα πρέπει να γίνει μια πολιτική συζήτηση για την διαιώνιση αν θέλετε και βελτίωση του συστήματος. Η ελεύθερη χορήγηση αδειών σημαίνει ότι θα υπάρξουν περισσότερα εισοδήματα για τα κράτη-μέλη και πιο δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων από το φόρο αυτό στο σύνολο των κρατών μελών. Εδώ είναι μια πολύ σημαντική πολιτική συζήτηση από την οποία νομίζω ότι θα εξαρτηθεί το μέλλον μας και στα πλαίσια του ETS αλλά και στον τομέα εκτός ETS. Τέλος, ο χρονισμός, το χρονοδιάγραμμα αν θέλετε. Είναι σαφές ότι αν προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή εξαρτώμεθα φυσικά και από τις προτάσεις της Επιτροπής Ήτρε δεν μπορώ να είμαι σαφής δηλαδή για το πώς θα εξαλειχθεί το χρονοδιάγραμμα, αλλά όπως είπα ο στόχος μου είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία στην Ολομέλεια του μηνός Ιουνίου για να είμαστε έτοιμοι πριν από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος τέλος Ιουνίου. Και ταυτόχρονα σαν Επιτροπή ΕΝΒΗ εμείς οργανώνουμε μία ακρόαση πάνω στο θέμα αυτό στις 28 Φεβρουαρίου ζητήθηκε να γίνει μια κοινή ακρόαση με την Ήτρε και την Έμβη, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε την χρονική πολυτέλεια να οργανώσουμε μια τέτοια συζήτηση και γι' αυτό ακριβώς με πραγματισμό αποφασίσαμε να κάνουμε μια ακρόαση το Φεβρουάριο, η Ήτρε θα κάνει τη δική της ακρόαση τον Μάρτιο, ελπίζω να καταλήξουμε σε μια εσωτερική ψηφοφορία στην Ήτρε στις αρχές Μαΐου και αρχές επίσης Μαΐου και σε μας για να φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Το θέμα είναι να ακούσω πολιτικά σχόλια. Τα δεδομένα τα ακούσαμε, τα επιχειρήματα τα ακούσαμε. Πρέπει να τα μετατρέψουμε σε πολιτικό λόγο. Περιμένω τις προτάσεις σας. Πρόεδρος Λάινενς, <clears throat> σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολλούς συγκεγραμμένους ομιλητές. Όπως είπα στην αρχή της συνεδρίασης, το πολύ δύο λεπτά, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Τονίζω και πάλι τη συνεργασία με την Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας. Είναι ένα θέμα όπου και οι δύο έχουμε αρμοδιότητες, άλλωστε και οι συνάδελφοί μας στη Ήτρε έχουν κληθεί να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί μας. Εγώ θα αναφέρω δύο μονάχα θέματα. Το να ανέβουμε στο 30% θα σημάνει ότι ορισμένες χώρες μέλη θα χρειαστεί να αγωνιστούν πολύ για την προσπάθεια αυτή, καθώς επίσης και ορισμένες βιομηχανίες. Νομίζω ότι είπατε και εσείς τα σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές και η Ιούτα Χάουκ η οποία ασχολείται στην Επιτροπή της ειδικά με το θέμα αυτό δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε όμως ειδικά τώρα θέματα κονδυλίων χωρίς να έχουμε την πιθανότητα χρηματοδότησης, διότι ορισμένε χώρες μέλη με επιβαρημένα ισοζύγια πληρωμών δεν θα ε, μπορέσουν να ανταποκριθούν ή τουλάχιστον θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές δυσχέρειες. Ήδη με το 20% ορισμένε χώρες μέλη καλούνται να αγωνιστούν ιδιαίτερα σκληρά. Για την βιομηχανία υπάρχει η πράσινη βιομηχανία η οποία αναζητά τρόπους αλλά έχετε και τις άλλες βιομηχανίες οι οποίες αγωνίζονται να επιβιώσουν στην παγκόσμια αγορά. Και ο τίτλος σας είναι «Ο κίνδυνος της λεγόμενης ε, ε, διαρροής άνθρακος» που πάει να πει δηλαδή τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές του κόσμου που είναι, όπου είναι ευνοϊκότερες οι ρυθμίσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ευφυής, ένας συνδυασμός πολιτικών να πιστούν εν τέλει όσοι δυσχεραίνονται να ε, προχωρήσουν. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και πρώτα στον κύριο Ταταρέλα. Εάν είναι παρόν. Καταρχάς, Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη συνεργασία, την το πνεύμα συνεργασίας το οποίο επέδειξε. Ραπόρτο. Ha ribadito anche oggi di avere molto έχει επανειλημμένα πει ότι είναι πράγματι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενος στο να βρεθεί μία λύση ε, και συνεργασία με την Ήτρε. Αλλά κάτι τέτοιο ίσως είναι ασύμβατο θα έλεγα με την ταχύτητα με την οποία θέλει να επεξεργαστούμε αυτήν την έκθεση. δεν μπορέσαμε καν να οργανώσουμε μία κοινή ακρόαση λόγω ακριβώς του ιδιαίτερα, της ιδιαίτερα πυκνής ημερήσιας διάταξης των εργασιών και των δύο επιτροπών. Εάν θέλουμε πράγματι να συνεργαστούμε για ένα καλό αποτέλεσμα, έχουμε κάθε συμφέρον η συνεργασία αυτή να ολοκληρωθεί και με μεγάλη πλειοψηφία βέβαια, δίδοντας σε όλους την δυνατότητα να εκφραστούν. Η ίδια έκφραση θα έλεγα και η ίδια προσπάθεια χρονική την οποία επιδεικνύει σήμερα ο εισηγητής σίγουρα μπορεί να αποδεί κάτι το χρήσιμο αλλά γνώμη μου προσωπική είναι ε, από μία πλευρά θα έλεγα τουλάχιστον. Αν υπάρχει μία παρουσίαση όλων των μελετών και όλων των συστημάτων τα οποία προτείνονται στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να πω εδώ ότι θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη η πρόταση του εισηγητή και να παρουσιάζει τις απόψεις ε, πληρέστερες, ευρύτερες, ε, γιατί μου φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εκφράζονται κάποιες πολύ συγκεκριμένες θέσεις, θέσεις όχι ιδιαίτερα ισόρροπες τα χαρακτήριζα. Επανερχόμενο σε αυτά τα οποία ακούστηκαν λοιπόν ο συνάδελφος μάλιστα Ζέμπερ, θα ήθελα εμείς, δεν έχω πια χρόνο, α, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Κοιτάξτε, έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα. και δίνω το λόγο στον κύριο Γιώργενσεν. Ευχαριστώ αυστηρά πρόεδρε. Θέλω να πω ότι το έγγραφο του εισηγητού είναι εξαιρετικό. Τον συγχαίρω λοιπόν. Λίγα λόγια τώρα σχετικά με τα διάφορα επιχειρήματά του. Πρώτα, ένα επιχείρημα που νομίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσει κύριε Σιγητά ακόμη περισσότερο, καθώς και στην ανακοίνωση και στη συζήτηση. Το γεγονός δηλαδή ότι ήδη έχουμε ήδη σχεδόν φτάσει στον στόχο του 20%. Πράγματι, ενδέχεται να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου λόγω των δυνατοτήτων αναβολής από το 2009 μέχρι το 2020 να δούμε αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του ανθρώπου Και φανταστείτε τι θα σημαίνει αυτό για τον πρωτοπόρο ηγετικό μας ρόλο ανά τον κόσμο. Ο μόνος τρόπος για να ασκήσει επιρροή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη soft power που διαθέτει με το καλό παράδειγμα δηλαδή. Η σωστή νομοθεσία είναι βέβαια καλό παράδειγμα, αλλά φανταστείτε εάν ξαφνικά βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου λόγω των διαφόρων offset οι ίδιες οι χώρες μας από το 9 και μετά αυξήσουν τις εκπομπές τους. Αυτό είναι πραγματικός κίνδυνος. Υφίσταται. Επίσης, αναφερθήκατε στην Κίνα ως καλό παράδειγμα. Και βρίσκω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ο Charles Friedman, αρθρογράφος του New York Times, έλεγε «Μακάρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ήταν Κίνα για μία μέρα». Και καταλαβαίνω τι εννοεί. Διότι αυτό που συμβαίνει σε αυτό το διαφορετικό βέβαια πολιτικό σύστημα τη Κίνα, είναι ότι πραγματικά προχωρεί με μεγάλη ταχύτητα προ τα εμπρό. και πράγματι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα αυτό διότι εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί με του ίδιου ρυθμού, θα μείνει πολύ πίσω στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Τέλο, συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να το ολοκληρώσουμε τον Ιούνιο την προσπάθεια αυτή ώστε να ε, προβαδίσουμε απέναντι και στα άλλα θεσμικά όργανα τηρήσατε τον χρόνο σας, ο κύριος Κρίς Ντέιβις. Είδα μια διαφήμιση για ένα αυτοκίνητο Fiat, ένα μικρό αυτοκίνητο, που παράγει 95 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακος ανά χιλιόμετρο. Αυτό για να μας δείξει πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει η τεχνολογία όταν θεσπίσει κανείς προδιαγραφές που την αναγκάζουν να προχωρήσει. Το ίδιο και οι αυξήσει βέβαια των τιμών των καυσίμων. Άρα υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει το δυναμικό. Έχετε την υποστήριξή μου για την έκθεση. Μπορείτε να το υπολογίσετε βέβαια αυτό. Γιατί και η ε, πολιτική της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στο 30% με την μεγαλύτερη, ε, με, στην πρώτη δυνατή ευκαιρία, όπως ε, άλλωστε την υποστηρίζει και ο γειτονάς μου από πίσω. αλλά ζούμε σε ένα πραγματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα πραγματικά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν στην έκθεση. Το πλαίσιο για να φτάσουμε στο 30% ήταν ότι θα υπάρχει μια διεθνή συμφωνία, άρα θα υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια συμφωνία. Ούτε υπάρχει πιθανότητα να εξασφαλιστεί υπογραφή τέτοια διεθνού συμφωνία για τα επόμενα χρόνια. Άρα, οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει αντιμετωπίζουν στην ουσία ένα δυσχερέ ανταγωνιστικό πλαίσιο με κίνδυνο ε, με κατάσταση επιχειρήσεων, ε, εξαγωγής της παραγωγής και εισαγωγής ε, ε, απασχόλησης και ούτω καθεξής. Άλλος παράγοντας είναι ότι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτό το 30% είναι με τα λεγόμενα offset. Αλλά ποια διάρθρωση θα ισχύσει για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που λέει ο εισηγητής μας Μπάζ λέει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε offset. Οι επιχειρήσει όμω βασίζονται σε αυτά, καθώς επίση είμαι βέβαιος ότι και η Κομισιόν. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για το μέλλον των offset αυτών. Α λάβουμε υπόψη λοιπόν τα αντίθετα επιχειρήματα όταν θα αξιολογήσουμε το περιεχόμενο τη έκθεση. Σα ευχαριστώ, Κρι, ο κ. Κάλαναν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχει κανένα νόημα να μιλήσω τώρα εγώ μετά από τον Chris Davis που ε, ήδη τα είπε αυτά που θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να κάνω λίγες παρατηρήσεις δικές μου. Πρώτα ευχαριστώ τον ε, φίλο μας Μπάς για μια έκθεση που προσφέρει τροφή για σκέψη όπως πάντα η εκθέση του έχει και ε, επιχειρήματα τα οποία αποτελούν πρόκληση για όλους μας για το ενδεχόμενο της αύξησης, της μείωσης δηλαδή στο 30%, εγώ πάντοτε ήμουν επιφυλακτικός κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο αυτό να πάμε το 20% στο 30%. Το κόστος το υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπου 81 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα εγώ υποθέτω ότι θα αποδειχθεί και πολύ υψηλότερο το κόστος αυτό. Πάντως αυτό είναι το επίσημο κόστος και διερωτώ με και για ποιο σκοπό εν τέλει ο Νταν Γιόργενσεν είπε ότι είναι σημαντικό να δώσουμε το καλό παράδειγμα, έστω το δέχομαι αυτό, δεν είμαι βέβαιος όμως ότι αναμένει αυτό το καλό παράδειγμα από εμάς ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Μπάς αναφέρεται και στην Κίνα. Οι Κινέζοι ναι, στέλνουν ενθαρρυντικά μηνύματα, βέβαια παράγουν πολλές αιωλικές γεννήτριες και μηχανήματα συλλογής της ηλιακής ενέργειας, αλλά κυρίως για να τα πουλήσουν σε εμάς δεν ξέρω εάν πραγματικά έχουν δεσμευτεί σε τίποτα για την ώρα. Έχουν τα πενταετή σχέδιά τους ή τα δεκαετή σχέδιά τους, όπως είπα, δίνουν κάποια θετικά μηνύματα, αλλά στις διεθνείς συζητήσεις δεν φάνηκε καμιά απολύτως διάθεση από πλευρά των Κινέζων, αλλά ούτε και από τους Αμερικανούς άλλωστε, να υπογράψουν κάποια δεσμευτική συμφωνία. Βέβαια, οι Κινέζοι είναι, για τους Κινέζους είναι σωστό μάλλον να κοιτάμε τι κάνουν παρά να ακούμε τι λένε και εγώ θα συμφωνούσα αν είναι δυνατόν με κάποια περαιτέρω μείωση, αλλά πρέπει να εξετάσουμε τα πραγματικά αποτελέσματα, τι πραγματικέ επιπτώσει. Πολλέ βιομηχανίε στην Ευρώπη μα λένε ότι ούτω ή άλλω δυσχεραίνονται πολύ να επιτύχουν έστω και το 20%. Εάν τώρα πρόκειται να τι εκδιώξουμε τον τρόπο αυτό για να φύγουν από την Ευρώπη να πάνε αλλού, δεν επιτυγχάνουμε τίποτα. Ήδη σε πολλού τομεί το ίχνος, όπως ε, για τη χαλιβουργία, την βιομηχανία αλουμινίου κλπ. Ναι, σας ευχαριστώ, πρέπει να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρος. Δυστυχώς συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά με διακοπτή Πρόεδρος. Λυπούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Οφείλω να σας ζητήσω να τηρήσετε τα όρια χρόνου. Η Σαμπίνε Ουίλς. Ευχαριστώ. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τον Μπάς τα επιχειρήματά του είναι ορθά. Η έκθεσή του δείχνει άλλωστε και την έλλειψη ασφάλειας που διέπει την ε, προσπάθεια, την πολιτική αυτή για την μείωση των διοξιδίων του άνθρακος. και στην προσπάθεια να τηρηθούν υψηλά οι τιμές των πιστοποιητικών για την εκπομπή διοξιδίων του άνθρακος και για να διατηρηθεί η, λειτουργία του μηχανισμού ε, ανταλλαγής κλπ. Τα 14 εκατομμύρια τα οποία έχουν, έχουν υπολογιστεί ότι θα είναι το όφελος από το ETS στην πρώτη φάση, στην πραγματικότητα καλύπτουν από πίσω το, το πρόβλημα ότι δηλαδή και για τις χώρες μέλη υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια σε ό,τι αφορά το σύστημα. Ο, ο Βάς λέει στην γνωμοδότησή του ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα για την ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας εφόσον υπάρξει το 30% το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Κριτικά ε, στέκεται η έκθεση απέναντι στα πιστοποιητικά της λεγόμενης καθαρής ανάπτυξης. Προτείνει ένα σύστημα πολλαπλασιαστών. Εγώ είμαι υπέρ να καταργηθεί το σύστημα CDM, το οποίο μάλιστα το οποίο μάλιστα έγινε κατάχρηση για να δικαιολογηθεί η παραπέρα χρηματοδότηση ανθρακοριχείων. Εγώ είμαι υπέρ μιας φιλόδοξης νομοθεσίας για την σωστή αποδοτικότητα της ενέργειας, το οποίο θα οδηγήσει και σε ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Rosbach. Tak, formand. Først tak til, til Bas. Det er et kolossalt arbejde, du har lavet. Det er et meget grundigt stykke papir, og jeg... Έχω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια τεράστια προσπάθεια έχει ήδη ε, διατυπώσει μια, ένα έγγραφο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο όμως παρουσιάζει και κάποια ανισχυτικά σημεία. Είναι αλήθεια ότι καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Διαρωτώ όμως αν υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι να διώξουμε την παραγωγική μας ε, δυναμική σε άλλες χώρες, στην Ινδία, παράδειγμα, νομίζω ότι κάθε Ευρωπαίος θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς καταναλώνει και γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα, να πληροφορήσουμε καλύτερα. Είναι κάτι το οποίο λείπει σήμερα. Όταν μιλάμε για τις οικοδομές, για τις κατοικίες και για την εξοικονόμηση ενέργειας, λίγα ακούγονται. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, λέει ο κ. Φλόρεντς, με την υπόδειξη ότι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Όπως το είπε εξής η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν οι χώρες μέλη εφήρμοζαν και αυτές μας οδήγησαν στην άθλια κατάσταση που βρισκόμαστε πολύ μακριά από το 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε ξεκάθαρη προσπάθεια να φτάσουμε στο 20%. Για τον παραδειγματικό χαρακτήρα των δράσεών μας βέβαια πρέπει να σημειώσω ότι θα πρέπει και να μπορούμε και σε αυτή την περίπτωση δεν το βλέπω. Είναι μια ενδιαφέρουσα απαρίθμηση διαφόρων φορέων ή παικτών που έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν για το κλίμα. Θα ήθελα πολύ να συμφωνήσω, αλλά η άποψη της βιομηχανίας και το ε, θέμα της ανταγωνιστικότητας. Αυτά δεν είναι παιχνιδάκια. Δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω για παράδειγμα μια χαλιβουργία. Και αν τη βγάλω απ' έξω τη χαλιβουργία, τότε η οικονομία ολόκληρη πάει πολύ άσχημα. Πρέπει να δούμε λοιπόν και από την άλλη πλευρά τι μπορούν να προσφέρουν οι οικονομικοί παίκτες, οι φορείς δηλαδή της οικονομίας και στο μέλλον να υπάρξει ενδεχομένως ένα ταμείο του προπολογισμού για την ε, αποδοτικότητα της ενέργειας. Ναι, αλλά αγαπητή Γιούτα, όπως ξέρεις, εκεί θα χρειαστεί να βάλει το χέρι πάλι στην τσέπη η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία για να πληρώσει τα χρήματα που θα πάνε στο Ταμείο αυτό. Η πολιτική της αποδοτικότητας στην οποία αναφέρθηκες αγαπητέ Μπάς, αυτή μου αρέσει πολύ είναι εκεί πραγματικά ένας τομέα όπου μπορεί να προκύψει και πράσινη απασχόληση και που ακόμα δεν έχει γίνει κατανοητό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυστυχώ. Το έγγραφο από τη μια μεριά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια μεριά των ενδιαφερόμενων, δηλαδή από την άλλη πλευρά των άλλων ενδιαφερόμενων, δηλαδή μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Αυτό που έχουμε ήδη εγκρίνει και σπανίως συμφωνώ με τον φίλο Κάλαχαν αλλά έχουμε συμφωνήσει 20% και 30% εάν συμφωνήσουν και άλλοι, αν υπάρξει διεθνή συμφωνία. Αυτό έχουμε αποφασίσει νομοθετικά και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, λέει ο Γιώ Λάινεν. Βέβαια και 30% δεν θα σήμαινε ότι θα επιστρέψουμε στην λίθινη εποχή, ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ορισμένοι έχουν εκφράσει την ε, τρομερή τους ανησυχία για το ότι θα, ε, υποτίθεται ότι θα σήμαινε. Θα τα συζητήσουμε αυτά βέβαια. Ο Ματίας, κοιτάξτε, για το πακέτο της ενέργειας έχουμε γκριν το 20% και αν συμφωνήσουν και άλλες χώρες το 30%. Φτιάξαμε και ένα ωραίο ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο, το οποίο δυστυχώς δεν έχει νομοθετικό περιεχόμενο. Σε θέματα άνθρακα τίποτα δεν έχει εγκριθεί νομοθετικά. Ένας στόχος του 2% έχει εγκριθεί. Και αυτό που δεν βλέπω στο ψήφισμα είναι ότι έχουμε, βρισκόμαστε μέσα σε μια οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Ναι, μείωση των εκπομπών. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να περάσουν ε, τα πιστοποιητικά στην επόμενη περίοδο από το 5% 8%. Άρα έχει μια ενδογενή αδυναμία το σύστημα. Χρειαζόμαστε μια ανάλυση και εδώ στο Κοινοβούλιο, εάν συμφωνήσουν και άλλοι παγκοσμίω για να φτάσουμε στο 30%. Και τότε οι μηχανισμοί που ήδη έχουμε εγκρινεί, για παράδειγμα ανανεώσιμες ενέργειες για το 2020 να φτάσουν στο 20%, ότι αυτό δεν θεμελιώνεται και με προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον και να υπάρξει και ένας μηχανισμός με πράσινα πιστοποιητικά, ένα ευρωπαϊκός μηχανισμός με πράσινα πιστοποιητικά. Και χώρες για τις οποίες συζητούμε, χώρες μέλη δηλαδή, βρίσκονται σε ε, ανανεώσιμε ενέργειε ακόμη πάρα πολύ πίσω. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα να φτάσουμε το 30% και μάλιστα με αποδεκτό κόστος. Διότι εν τέλει την ύφη θα την πληρώσουν οι πολίτες. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιστρέψουμε την ε, πολιτική του κλίματος και να δούμε εάν κάποιοι θα δεχθούν να μας ακολουθήσουν από τον υπόλοιπο κόσμο και με φιλόδοξα ποσοστά να είχαμε πάει στο Κανκούν και με 40 και με 50% μείωση να είχαμε πάει στο Κανκούν δεν νομίζω να είχαμε εντυπωσιάσει κανέναν. Θα πρέπει αντίθετα να είμαστε έτοιμοι αν τελικά προκύψει διεθνή δεσμευτική συμφωνία να μπορούμε να μειώσουμε στο επίπεδο 30%. Αν άλλοι δεν συμφωνήσουν τότε να προσπαθήσουμε να φτάσουμε το 20%. Υπενθυμίζω την ανάγκη των 20 λεπτών γιατί έχουμε ακόμα το θέμα της διοξίνης καθώ και πολλά άλλα θέματα. Περιμένουν ήδη απ' έξω οι συνομιλητές μας. Θα σας πω τώρα ποιοι είναι οι επόμενοι. Τώρα επόμενος είναι ο κύριος Αρσένης. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την τεράστια δουλειά που έχεις κάνει, πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο και τα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνει εντυπωσιάζουν. Ποιο είναι το κόστος λοιπόν του 30%? 70 δις περίπου. Έτσι φέρεται 11 μάλλον δις, ενώ 50 δις είναι το κόστος ε, αντιμετώπισης ε, των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν μετά το 2011. ιδιαίτερα σχετικά με το κόστος που θα προέλθει από τη φορολόγηση του μη ETS τομέα. Τι σημαίνει αυτό. Το κόστος αυτό νομίζω μπορεί να καλυφθεί πληρώνοντας μόνο για κάθε θέση εργασίας που θα δημιουργηθεί 11.000 ευρώ. Πολύ συχνά αυτό μας κοστίζει πολύ περισσότερο. Θα πρέπει να δούμε βέβαια να μην ξεφύγουμε. Ξέρουμε ότι το κόστος αυτό αντίστοιχα θα είναι υψηλότερο στο μέλλον. Η κλιματολογική αλλαγή δεν είναι της μόδας απλά, δεν είναι μια τάση είναι μια πραγματική απειλή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε μέτρα. Το θέμα είναι πότε θα τα πάρουμε τα μέτρα αυτά. Για την Κίνα, παρότι αποτύχαμε στην, αποτύχαμε στην Κοπενχάγη, η Κίνα κάνει τη δική της δουλειά με δικούς της στόχους, είναι σαφές ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ποσοστά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των κλιματολογικών αλλαγών και αν δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Κίνα σήμερα, πώς θα το κάνουμε με μια πράσινη Κίνα στο μέλλον. Λεπάζ. Συμφωνώ με τον συναδέλφους και συγχαίρω τον εισηγητή. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίασή του. Θα είμαι πολύ σύντομη να υπογραμμίσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο οικολογικό και καταπολέμηση των συνεπειών της των κλιματολογικών αλλαγών. Είναι βιομηχανικό πρόβλημα, είναι θέμα βιομηχανικών συγκρούσεων. Μετά τον Κανκούν υπήρξε θα έλεγα μια γρήγορη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις χώρες του Νότου και κατά συνέπεια σε πολιτικό, γεωστρατηγικό και οικονομικό επίπεδο αν η Ευρώπη δεν επενδύσει μαζικά στον τομέα αυτό τότε είναι σαφές ότι θα χάσουμε κάθε ηγετική προσδοκία και φιλοδοξία στον οικονομικό τομέα. Συνεπώς λοιπόν οι επενδύσεις τις οποίες θα κάνουμε τώρα θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την οικονομική μας εξέλιξη τα επόμενα δέκα χρόνια. Αν χάσουμε το τρένο τότε δεν θα ξαναπεράσει το επόμενο δρομολόγιο. Λοιπόν, το να βάλουμε υποχρεώσεις σε επίπεδο εσωτερικό μονομερές στην ουσία είναι σαν να αντιπάρουμε τη βιομηχανία μας. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γνωρίζω τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας τα οποία αναφέρθηκε ο Φλόρενς και άλλοι, αλλά δεν έχουμε όμως άλλη δυνατότητα. Η Βραζιλία, το Μεξικό, η Κίνα, η Ινδία ακολουθούν την κατεύθυνση αυτή και δεν μπορούμε εμείς να μείνουμε πίσω. Merci beaucoup, ο κ. Ζέμπερ, ευχαριστώ και εγώ τον Μπάς με τη σειρά μου για το έγγραφό του καθώς και για την διάθεσή του να οργανώσει ακρόαση μαζί με την Ήτρε. Το θεωρώ σκόπιμο. Βέβαια, το έγγραφο μου προκαλεί ορισμένα προβλήματα και κυρίως ό,τι αφορά τα νούμερα που από άλλα Ινστιτούτα το κόστος που ε, εμφανίζουν είναι πολύ υψηλότερο, καθώς επίσης και η βιομηχανία που έρχεται και μας βλέπει θεωρεί ότι χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις στα νούμερα. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι μια έλλειψη συνέχειας. Λέει στο έγγραφό του ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα κλπ. είναι πολύ πιο προχωρημένες από, εδώ, από ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη και όμως αυτές οι χώρες είναι οι οποίες είναι τόσο έντονα αντίθετες με οποιαδήποτε δεσμευτική διεθνή συμφωνία. Διαρωτώ με μήπως εμείς είμαστε στο σωστό δρόμο, οι Ευρωπαίοι δηλαδή και το περίφημο ETS και το burden sharing είναι η σωστή προσέγγιση ή μήπως άλλες χώρες οι οποίες μάλιστα εκπέμπουν περισσότερο διοξίδιο άνθρακα τα καταφέρουν καλύτερα δίνοντας διαφορετικά και καλύτερα κίνητρα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα, πολιτικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Δηλαδή πώς από τη μια μεριά θα είμαστε επιτυχημένοι σε ό,τι αφορά την προσπάθεια μείωση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και ταυτόχρονα μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα μέλλον εδώ στην Ευρώπη. Με την προσέγγιση του, αυτή τη γραμμική δηλαδή προσέγγιση προς το 30% νομίζω ότι είναι εσφαλμένος ο δρόμος αυτός. Και η πολιτική μου ομάδα νομίζω έχει την ίδια γνώμη μαζί μου και γι' αυτό θα θεωρήσει ότι χρειάζονται κάποια τροποποίηση για τα ETS 50% εκτός Ευρώπης, για το burden sharing 80%. Πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε ωστόσο να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις. Για την ιδέα τώρα, περιφερειακή πολιτική και αγροτική πολιτική να ενταχθούν μέσα σε μια περιβαλλοντική πολιτική, συμφωνώ. Αλλά προσοχή, οι συνάδελφοί μας της ε, Επιτροπής Γεωργίας έχουν διαφορετική άποψη. Θα χρειαστεί λοιπόν να μην κάνουμε το λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Πρέπει να, ε, πρώτα να συζητήσουμε μαζί τους. Ευχαριστώ. Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούστηκαν πάρα πολλά και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας να πω ότι συμφωνώ βεβαίως με αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής Μαζέμπερ σχετικά με τους αριθμούς. Νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, να είμαστε πιο σίγουροι και περισσότερες διαφρυνήσεις σχετικά με τις προτάσεις τις οποίες κάνει. Γιατί υπάρχουν κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι αντίθετα με συμπεράσματα άλλων μελετών και ερευνών. Εν πάση περιπτώσει μπορεί κανείς να διαφωνεί πάνω στους αριθμούς όταν σαν παράδειγμα λέγεται ότι η αύξηση του κόστους για να περάσουμε από το μείον 20% στο μείον 30% θα είναι γύρω στο 16% ε, ναι, 16% ε, πάνω στις προβλέψεις που είχαν γίνει για τη μείωση του σε 20% του 2008, ενώ πρέπει να δούμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα σήμερα, το 2011 και γι' αυτό θα μπορούσε να υπάρξει μια αναπροσαρμογή θα έλεγα των υπολογισμών και των στοιχείων για να δούμε τι θα κάνουμε με τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αν βασιστώ στο κόστος που έχει υπολογιστεί το 2010 βλέπω ότι η αύξηση δεν είναι 16% αλλά 69%. Μιλάμε για μια τεράστια διάσταση. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πιο σίγουροι με τα ποσοστά και τους αριθμούς όταν αντιπαρατήθεμεθα και νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο και να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Βλέπω ότι και η ΕΕ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λέγει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα αν λειτουργήσει αυτόνομα και αν και οι εταίροι μας δεν πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις και αν δεν υπάρξουν ιδιαίτεροι προστατευτικοί δασμοί τότε θα οδηγηθούμε σε μετακινήσεις επιχειρήσεων πάρα πολύ σημαντικές. Ξέρουμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια μας κοστίζει 20% περισσότερο από τις Ηνωμένε Πολιτείες και 25% περισσότερο από την Κίνα. Όλα αυτά θα χειροτερεύσουν στο μέλλον. Eh, Κυρία Γκοστέτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ακούστηκαν, θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω την επιφυλακτικότητα την οποία είχα πάντα θα έλεγα εγώ πάνω σε ένα τέτοιο θέμα συγχαίροντας τον εισηγήτη γιατί η έκθεσή του τουλάχιστον προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον αν μη τι άλλο. Όπως σας είπα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί το λέω αυτό. Πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, όταν αναφερόμαστε στην Κίνα, αυτό το οποίο φοβάμαι είναι ότι η Κίνα έχει καταλάβει ότι θα πρέπει να αναπτύξει καθαρές τεχνολογίες για να κατακτήσει για μια ακόμη φορά την ευρωπαϊκή αγορά και να ανταγωνιστεί τις επιχειρήσεις μας. Και εν τω μεταξύ η Κίνα συνεχίζει να εγκαινιάζει δεκάδες μονάδες παραγωγής με άνθρακα. Συνεπώς υπάρχει εδώ ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Κίνα έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι η αγορά είναι ενιαία, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσα σε αυτή την αγορά για να ανταγωνιστεί και να κατακτήσει τη δική μας εσωτερική αγορά. Συμφωνώ επίσης με την Κορίν Λεπάζο όταν λέγει ότι η συζήτηση δεν είναι μόνο οικολογική αλλά και οικονομική. Βεβαίως όταν μιλάμε για βιομηχανική πολιτική εννοείται Ας κάνουμε λοιπόν κάποιες προσπάθειες και σε έναν τομέα μπορούμε να δράσουμε, είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή όμως, όχι μόνο οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες και τίθεται εδώ το θέμα του προϋπολογισμού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε εμείς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ένας είναι ο κανόνας, πρέπει να επιβληθεί σε όλους, είναι ο κανόνας της αμοιβαιότητας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας λοιπόν. Ήταν, θυμίζω, η πρώτη συζήτηση γύρω από το έγγραφο εργασίας. Ε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην φάση της έκθεσης. Στι 28 Φεβρουαρίου θα έχουμε μια κρόαση μέσα στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Ένα πρωί θα είναι ή απόγευμα, όπου θα έχουμε χρόνο, τρει ώρες πάλι, ώστε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Και μετά στις 16 Μαρτίου, όταν θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης και θα το συζητήσουμε, και εμεί λέμε ότι στις 22 Μαρτίου θα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών η έκθεση πιο πριν θα είναι φυσικά στη διάθεσή σας. Το Μάιο, αν γίνεται, θέλουμε να ψηφίσουμε προς έγκριση, ώστε τον Ιούνιο να περάσει στην Ολομέλεια. Αυτό είναι, ας το πω έτσι, το ευκταίο χρονοδιάγραμμα. Αν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ήτρε τα καταφέρουν πριν από την Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, θα είναι καλό να έχουμε την έκθεση. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την εκκίνηση αυτής της συζήτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ θερμά με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά, συμφωνώ, πολλά διακυβεύονται και το ένα και το άλλο για την προστασία του κλίματος αλλά και για τη βιομηχανία, την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ακούστηκαν τα επιχειρήματα, ωραία. Τώρα, μια και πιέζει ο χρόνος, προτείνω να περάσουμε στο επόμενο μείζον θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Πράγμα το οποίο αφορά την ασφάλεια τροφίμων. Και πριν από την ασφάλεια τροφίμων και μετά ε, τις ζωοτροφές που καταναλώνουν τα ζώα στην κτηνοτροφία. Το σημείο 12 στην ημερησία διάταξη είναι το θέμα της διοξίνης και της μόλυνσης με διοξίνες των ζωοτροφών. Εδώ υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε και που έχει ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα στις επιπτώσεις του. Έχουμε το Europe by Satellite ανάμεσά μας, τη δική μας τηλεοπτική ομάδα, τον σταθμό μας που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα Επίσης έχουμε και την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, Πάολα Χριστόρη. Καλώς ήρθατε, θερμό καλώς ορίσατε. Και θέλουμε να ξέρουμε από εσά και το ζήτησε και η κυρία Ροτ αλλά και άλλοι να το ακούσουμε, τι σκοπεύει να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν οι ελλείψεις που ε, σημειώθηκαν και διαπιστώθηκαν και σήμερα έχουμε τους Υπουργούς ε, <clears throat> Γεωργίας στις Βρυξέλλες που συνεδριάζουν και διαβουλεύονται για αυτό το θέμα, συσκέπτονται γι' αυτό. Νομίζω έγκαιρα και <clears throat> σε σωστή χρονική στιγμή ασχολείται η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τους αδύναμους κρίκους για την τροφική αλυσίδα, την ασφάλεια τροφίμων. λάβει... Α, δεν ήταν το έτοιμά σας να παρέμβετε εσείς κύριε Εντάξει, τότε η τα και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να αποχωρήσω. Έχω παράλληλα ανηλυμένες υποχρεώσεις, αλλά θα αναλάβετε εσείς την Προεδρία τη απουσία μου. Κύριε Βεστόρη, έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι πράγματι το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας ε, συζητά αυτό το θέμα, το συζήτησε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί. Είμαι επίσης σε θέση να σας πω ότι για αυτή τη συζήτηση να σας αναφέρω κάποια πράγματα και τα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι Υπουργοί, ότι το σύστημα ασφάλειας τροφίμων είναι λοιπόν σε σχέση με την ασφάλεια όταν σημειώνεται μια κατεπίγουσα, ένα κατεπήγον περιστατικό σαν αυτό, το σύστημα λειτουργεί, λειτουργήσε το σύστημα και για τη σταθερότητα όταν είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε μια μόλυνση μπορούμε να απομονώσουμε όλες τις ε, δυνάμει μολυσμένες αυτές τις κτηνοτροφικές μονάδες και παραγωγούς ζωοτροφών. Και σε πραγματικό χρόνο μπορέσαμε να διαδώσουμε, να διαχύσουμε τις πληροφορίες σε όλα τα κράτη-μέλη μέσω του συστήματος ε, άμεσης ε, προειδοποίησης. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτή την περίπτωση, για αυτή τη μόλυνση δεν υπήρξε άμεσα κίνδυνος υγείας. Γιατί εδώ κάνουμε λόγο για μια κατάσταση όπου το όριο διοξινών έχει ναι μεν ξεπεραστεί, αλλά το ξεπέρασαν μόνο κατά ελάχιστη ποσότητα. Κάνουμε λόγο για περιπτώσεις όπου κατά 1,5 ή 2 έχει υπερβεί, έχουν υπερβεί αυτό το όριο που δεν έχει κανένα σύγκριση με προηγούμενες παλαιότερες κρίσεις διοξίνης όπως ε, αυτές που σημειώθηκαν στην Ιρλανδία πριν από δύο χρόνια που είχαμε 200 πλάσια, 200 φορές ε, το όριο ή στο Βέλγιο το 99 που είχαμε χίλια πλάσιο όριο που είχαμε υπερ, είχαν υπερβεί. Έτσι λοιπόν ε, σε σχέση με τη, την μόλυνση ήταν ελάχιστη ε, στο σημείο υπέρβασης. Πολύ θετικά λοιπόν υπήρξε αντίδραση από πράσους ε, των Υπουργών για την Επιτροπή μας. Είπαν ότι σε μια τέτοια περίπτωση ε, έκτακτη ανά... έκτακτης ανάγκης πρέπει να συναγάγουμε κάποια μαθήματα. Πρώτο μάθημα, πρέπει απόλυτα να εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι νόμοι για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Είναι ένα πρόβλημα συμμόρφωσης και επιβολής ε, του νομοθετικού πλαισίου. Και ο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα, δηλαδή που έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη, εις βάρος όλων των κρατών μελών. Γιατί τώρα αυτό το κατεπήγον είχε επιπτώσει σε όλη την τροφική αλυσίδα της στην Ευρώπη. Είναι όμως σαφές ότι εμείς τώρα δεν προβληματιζόμαστε και δεν σκεφτόμαστε νέα μέτρα γιατί υπό όρους διοξίνης έχουμε ένα καλό σύστημα εποπτείας. Όλα τα όρια είναι καθορισμένα και το σύστημα ελέγχων υφίσταται. Αλλά υπάρχουν κάποια λίγα πράγματα που μπορούμε να πράξουμε για να γίνει πιο σφιχτό, πιο αποτελεσματικό και ασφαλές το σύστημα αυτό. Και η δική μου επιτροπή έχει προτείνει τέσσερα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εμείς στοχεύουμε να προτείνουμε και για τη μόνιμη επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες. Τα τέσσερα αυτά μέτρα είναι πρώτον, θεωρούμε ότι ο ε, παραγωγός σε σχέση με την ε, ε, επεξεργασία λοιπόν και κορεσμένων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη υποπτία. Εδώ υπάρχει αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα και πρέπει να εγκρίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Ενώ μέχρι σήμερα μόνο καταχωρούν σε κάποια μητρώα. Αυτή η παραγωγή λίπους θα πρέπει να μπορούν να παράγουν λίπος για, τεχνικούς, για τεχνικές χρήσεις αλλά και για ζωοτροφές. Είναι αναμεμειγμένο το πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Τώρα πιστεύουμε ότι πρέπει να, να υπάρχει μια ξεχωριστή παραγωγή. Είτε μέσω ξεχωριστής παραγωγής μέσω μονάδων, είτε διαχωρισμού των ίδιων των μονάδων παραγωγής. Να μην υπάρχει δυνατότητα μόλυνσης ε, από την τεχνική επεξεργασία για, την, ε, για τον τρόπο παραγωγής ε, των λοιπών. Όσον αφορά την εποπτεία διοξινών, δεύτερον, θέλουμε να εισαχθεί ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο συλλογή και αξιολόγηση τέτοιων κρίσιμων υλικών, κέριων υλικών όπω των λοιπών. Το λίπο, τα λίπη είναι κέρια στοιχεία και γι' αυτό πρέπει λοιπόν και δειγματοληπτικά να συλλέγονται και να αναλύονται. Και γενικά θα μεριμνήσουμε όλα τα στοιχεία τη εποπτεία διοξινών που υφίστανται ήδη να τα εκμεταλλευόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία σε, πλήρη, σε πλήρες μέτρο. Τέταρτο μέτρο που θέλουμε να εισαγάγουμε είναι θέλουμε να επιβάλλουμε στα ε, ε, ε, εργαστήρια την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα άμεσα όλες τις, όλα τα θετικά ευρήματα. Αυτή η υποχρέωση υποβολής αναφοράς. Οποιαδήποτε φορά σημειώνεται κάποια μόλυνση, τώρα θα είναι και για τους παραγωγούς τροφίμων και ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει για τους παραγωγούς τροφίμων και ζωοτροφών, αλλά όχι για τα εργαστήρια. Θέλουμε να επεκτείνουμε το εύρος αυτής, αυτού του κανόνα, αυτής της ε, ε ρύθμισης και για τα εργαστήρια. Και έτσι μέσω επιτροπολογίας είναι μικρές τροποποιήσεις και προσαρμογές αυτά. Δεν είναι νέα μέτρα, είναι ίσονος, ε, ας το πω έτσι, προσαρμογής ε, νέες, πρωτοβουλίας, νέες πρωτοβουλίες. Και θέλουμε στο πλαίσιο αυτό να εφαρμόζονται και να ελέγχονται αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ. Και ήταν πραγματικά μια έκπληξη αυτό το οποίο αναφέρθηκε για μένα. Έκπληξη για όσα είχαν συμβεί. Μπορούμε να αναμείνουμε Αυτά τα πράγματα δεν ξέρουμε αν θα συμβούν ή όχι πάλι πότε. Σε τρία, πέντε χρόνια δεν μπορούμε να μαντεύσουμε. Ε, στην Ιρλανδία ήταν χειρότερα, είπε στο Βέλγιο ακόμα χειρότερα από ό,τι στην Ιρλανδία και ο λόγος ήταν ο ίδιος. Έχουμε υπερβολική θέρμανση από ε, τις ε, μονάδες αυτές και αυτό, απέρευσε, αυτό οδήγησε σε αυτή τη μόλυση. Όταν άκουσα για πρώτη φορά στη Γερμανία το τι συνέβη, δεν ήξερα να, χαμα, να ή να αρχίσω να κραυγάζω για μια ανακοίνωση τύπου ε, σκέφτηκα, ορίστε, είχαμε 10, 15, πόσα, 20 τα τελευταία χρόνια με τον ίδιο τρόπο κιόλα, θέλω να υπογραμμίσω ότι όλη η νομοθεσία για τον έλεγχο τροφίμων και ζωοτροφών του 2004 είναι πολύ σύγχρονη νομοθεσία και πολύ καλή. Το πρόβλημα όμω είναι ότι δεν υλοποιείται, δεν εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Αν λέγατε στη Γερμανία ή ρωτούσατε τη Γερμανία άλλα κράτη, ποιο εποπτεύει και ελέγχει τι και τότε πραγματικά σε αυτό το επίπεδο, και το έχουμε πει πολλές φορές, ισχύει αυτό. Είναι πολύ σύγχρονη νομοθεσία. Δεν είναι ξεπερασμένη και ανεδαφική. Δεν ήταν λοιπόν κάποια ξεχωριστή δράση που να απαιτείται από τους Υπουργούς ε, Γεωργίας εκείνο που ζητούσαν ήταν να υπάρξει μια αλλαγή ε, στην ίδια το, στο ίδιο το πεδίο ευθύνη του γιατί πίστευαν ότι αυτό θα του ε, βοηθούσε. Θα μπορούσε από πλευρά ε, Γερμανία να είχε γίνει κάτι για παράδειγμα σε σχέση με τι ζωοτροφέ και τα τρόφιμα. Είναι αρμοδιότητα των κρατηδίων στη Γερμανία. Θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ίσω το κράτο θα μπορούσε κεντρικά να τα ρυθμίζει αυτά. Αλλά είναι διαφορετική η κατάσταση. Η υποχρεωτική βελτίωση τη αντιμετώπιση των λοιπών και των οξέων. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό. Δεν είχαμε πει όταν τότε υπήρχε η κρίση της σπογγόδους εγκεφαλοπάθειας των βοηδών ότι θα χρειαζόταν η έγκριση όλων των ε, παραγωγών εταιριών και δεν υπήρξε άμεσα αντίδραση και διαμαρτυρία μεταξύ των Υπουργών Γεωργίας και των παραγωγών ταυτόχρονα αντέδρασαν και είπαν πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει, πώς μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Ναι, εγώ σας υποστηρίζω, πρέπει να γίνει αυτό όμως. Πρέπει να είναι σαφής η ευθύνη εκείνο που παράγει τρόφιμα ζωοτροφές Είναι το πρώτο σκέλος στην αλυσίδα ε, της ε, ευθύνης. Να υπάρχει υποχρεωτική τέτοια αδειοδότηση και να θα είμαστε αρκετά θαραλέοι ώστε να εφαρμοστεί αυτό απόλυτα. Να είμαστε θαραλέοι και γενναίοι. Παρακαλώ, α είμαστε θαραλέοι. Υποχρεωτική εφαρμογή και έγκριση. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, τώρα μόνο σε, στην περίπτωση αυτή τη ε, όξυνση τη κρίση μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα δεν αλλάζει τίποτα βέβαια. Εγώ θα προτιμούσα αν παραμέναμε πιστοί στην ε, εφαρμογή σε συγκεκριμένα στοιχεία για την ε, ΣΕΒ της πογκώδη εγκεφαλοπάθειας στο παρελθόν που έπρεπε να ε, ρυθμιστούν ή να καταλήγουν στα απόβλητα και υπήρξε δυνατότητα χρωματισμού και αυτό ήταν μια καλή ιδέα Τώρα, για το άλλο το οποίο είπατε, όχι νέα μέτρα. Υποστηρίζω και εγώ ότι δεν χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Όμω αυτό που θα σα ρωτούσα είναι, μπορείτε να μα πείτε ίσω σήμερα κιόλα πώς τα κράτη-μέλη θα ανταποκριθούν σε σχέση με την υποβολή αναφορών, σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους, ε, σε σχέση με την νομοθεσία του 2004. Ποιοι είναι οι καλοί, τα καλά παιδιά και ποιοι τα κακά παιδιά. Και πόσο συχνά υποβάλλουν τέτοιες αναφορές. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα τα κράτη-μέλη να υποχρεούνται σε συγκεκριμένα προβλήματα που είχαμε, όπως τις διοξίνες, να τα υποχρεώνουμε να μετρούν το επίπεδο διοξινών γιατί για τα, από την νομοθεσία 2004 αφήνεται στα κράτη-μέλη να κρίνουν τι θα ελέγχουν και σε ποιο βαθμό και εύρος. Και τελευταίο στοιχείο, τελευταίο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω, πέρα από τα υπόλοιπα στα οποία σας υποστηρίζω, θα πρέπει να πω με ταπεινότητα και στρέφομαι προς τον συνάδελφο Στίβενσον που ίσως και δεν, θα, δεν προσέχει και τόσο πολύ. Θέλετε και πάλι να ε, ξαναδούμε τα όρια για τη διοξίνη στα μέτρα επιτροπολογίας. Ε, πώς λέγεται αυτό στα αγγλικά η ορολογία. Δηλαδή ανεπιθύμητες ουσίες στις ε, ζωοτροφές, στην κτηνοτροφία, στην διατροφή των ζώων. Θέλετε ξανά να τα ξαναδούμε αυτά σε σχέση με τα ηχθιάλευρα, για παράδειγμα, το επίπεδο διοξινών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι τα προτινόμενα μέτρα είναι στην σωστή κατεύθυνση και βέβαια καλούνται οι χώρες μέλη ανεξαρτήτως εσωτερικών διαμαχών περί της αρμοδιότητες να εφαρμόσουν τα όσα αποφασίζονται και εγκρίνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως, ο χωρισμός μεταξύ τεχνικών λοιπόν για την παραγωγή τροφίμων. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Θα μειωθούν και οι κίνδυνοι εάν ξεχωριστούν οι δύο διαδικασίες. Επομένως η πρόληψη θα βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες μολύνσεις. Και θα πρέπει να γίνονται και οι δοκιμασίες αυτές από όλους τους παραγωγούς και θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεχωριστό σύστημα ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ανιχνευσιμότητα. Ότι λειτουργεί το είδαμε, αποδείχθηκε, αλλά κάποιες βελτιώσεις απαιτούνται. Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης κατά πόσον μπορεί να βελτιωθεί μέσα στην ίδια την αλυσίδα η επικοινωνία. Να υπάρξουν πλατφόρμες δηλαδή όπου γίνεται επικοινωνία μεταξύ εργαστηρίων παραγωγής και χρηστών, μέτρο το οποίο θα συμβάλλει στην μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα στον τομέα και επομένως και στη μεγαλύτερη ασφάλεια. Και η αρχή που λέγεται στα αγγλικά name and shame, δηλαδή να ανακοινώνεται τα ονόματα των παραβατών, θα μπορούσε μάλιστα να γίνει αυτό στο διαδίκτυο ώστε να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές και είμαι πεπισμένη ότι η παραγωγή εκείνη ζωοτροφών που εργάζονται σωστά θα ωφεληθούν εν τέλει από ένα τέτοιο σύστημα. Και βεβαίως και ο καταναλωτής να γνωρίζει από ποιον αγοράζει και τι αγοράζει. Ένα μικρό πρόβλημα ερίστον παρόδο, μία ερώτηση, έχει εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν υπάρχουν διαδικασίες όπου μπορούν να προκύψουν τοξικές ουσίες από εσωτερικές χημικές αντιδράσεις για παράδειγμα για την παραγωγή βιολογικού ντίζελ ή λοιπόν από ε, φυτική βάση μπορεί να προκύψουν προσμένες διαδικασίες τοξίνες. Θα ήθελα να μάθω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχει κάποια, κάποια καινούργια αποτελέσματα έρευνας εν προκειμένου. Ευχαριστώ. Ο Κρήτον. Θα ήθελα να καταλάβω ποιες είναι οι δυσκολίες που εμποδίζουν ε, τα ατυχήματα αυτά να μην ξανασυμβούν. Έχουμε χώρες με καλά συστήματα για την αξιολόγηση και παρακολούθηση τέτοιων κινδύνων. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε να ξεσπούν κάθε τόσο πολλές ε, κρίσεις σε αναπτυγμένες ε, χώρες με αναπτυγμένα νομοθετικά πλαίσια. Όπως είπε και η Ντάκμαρ λοιπόν, δεν ξέρω αν ένα τέτοιο ατύχημα μπορούμε να το αποφύγουμε στο μέλλον. Από ό,τι φαίνεται, η διαδικασία παραγωγής τροφίμων είναι ανεξέλεγκτη. Και αυτό θα μας κάνει σύντομα θα έλεγα να βελτιώσουμε την παραγωγή, να προωθήσουμε την οργανική παραγωγή και να ακολουθήσουμε πρακτικές οι οποίες να μην είναι βλαπτικές για τη φύση. Πρέπει να το σκεφτούμε και εδώ και στην Επιτροπή αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Κλάης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την αναφορά σας. Ένα πράγμα με ενόχλησε βέβαια σε αυτά που είπατε. Ήταν βέβαια μικρή η ποσότητα, ήταν και μικρή η μόλυνση, αλλά απάτη υπήρξε. Αυτό είναι γεγονός. Και εκεί χρειάζεται να επιβληθούν κυρώσεις. Γιατί μόνο με κυρώσεις μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν οι απάτες αυτές. Έτσι είναι. Ορισμένοι λένε τώρα ότι οι ζωοτροφές είναι υπερβολικά φτηνές, αλλά και ακριβότερες να ήταν, πάλι θα γινόντουσαν απάτες, γιατί τότε και το περιθώριο κέρδους θα ήταν μεγαλύτερο. Οι χωρισμένοι μέλη οφείλουν να φροντίσουν και βεβαίω η ε, δική μας υπουργό θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Τα επιχειρήματα προβλήθηκαν ότι δεν είναι και σύνηθες κάτι τέτοιο, ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αναφορές όταν διαπιστώνουν κάποια ε, αξιοσημείωτα περιστατικά. Αυτό πρέπει να γίνεται όμως για να μην επαναληφθούν τέτοια πράγματα. Το ότι πρέπει να εξετάζονται οι ζωοτροφές το βλέπουμε. Δεν είναι δυνατόν να μην ε, υπάρξουν διαρκείς έλεγχοι το κρασί που πωλείται κάθε παρτίδα ε, κρασιού εξετάζεται από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο. Το ίδιο πρέπει και για τις ζωοτροφές. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, για παρτίδες πάνω από 200 τόνους, γίνεται αυτομάτως εξέταση εάν υπάρχουν υπόλοιπα ε, κατάλοιπα τέτοιων ουσιών. Θα ρωτήσω λοιπόν τι γίνεται στο Βέλγιο τι αποδίδει η προσπάθεια αυτή. Είναι επιτυχημένη ή όχι. Βέβαια 200 τόνοι είναι πάλι πάρα πολύ από την άλλη μεριά. Θα πρέπει λοιπόν να οριστούν καλύτερα οι έλεγχοι και οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται και να δείξει το σωστό δρόμο η Ευρώπη. Επίσης, οι αγρότες οι οποίοι τώρα έχουν στους τάβλους τους ζώα τα οποία είναι σε ηλικία προσφαγή αλλά δεν μπορούν να τα απολύσουν τώρα είναι όμοιροι της επιχείρησης ζωοτροφών, της αλυσίδας παραγωγής ζωοτροφών. Δεν μπορούν όλοι οι αγρότες βέβαια να παράγουν τις ζωοτροφές στα αγροκτήματά τους για να ταΐσουν τα ζώα τους. Άρα είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν σωστές ζωοτροφές. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα καταστήσουμε δυνατό και στους αγρότες μας να παράγουν στο μέλλον καλής ποιότητας κρέας και ασφαλές για την κατανάλωση. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ η επόμενη ομιλήτρια να περιοριστεί στα δύο λεπτά για να προλάβουμε. Το... Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το σημερινό σκάνδαλο διοξινών αν είχαν γίνει κάποιες ε, εξετάσεις ε, και αναλύσεις προτού αναμειχθούν αυτές οι ουσίες με τις ζωοτροφές. Τότε η επιβάρηση θα είχε έγκαιρα διαπιστωθεί. Η παραγωγή ζωοτροφών πρέπει να υποχρεούνται κάθε οποιαδήποτε τέτοια ε, ουσία να την ελέγχουν προτού αναμειχθεί με ζωοτροφές. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κλάσσα διότι διαφορετικά δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα. Δεν μπορεί ούτε μία ουσία να εισαχθεί στις ζωοτροφές που δεν τηρεί τα όρια και όποιοι δεν τηρεί το όριο θα πρέπει να καταστρέφεται. Και τα μέτρα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι είναι σκόπιμα η νομοθεσία, οι νόμοι προβλέπουν ήδη σήμερα ότι αν οι οριακές τιμές δεν, δεν γίνεται μέσω ε, αποδυνάμωσης ή αρέωσης ε, να τηρηθούν, ε, πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές οπωσδήποτε. Είδαμε σε σχέση με τη βιομηχανία την ε, σημαντική αυτή μείωση και ότι η προσοντούχοι συνάδελφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και πρέπει ένα αντίστοιχο σύστημα ελέγχων να οικοδομηθεί, να δομηθεί. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα καταφέρει τα κράτη-μέλη να οδηγηθούν να συμμορφωθούν με αυτό. Ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει το σύστημα πιο ασφαλές. Θέλω να αμφισβητήσω ένα μέρος του συστήματος, την μαζική κτηνοτροφία δηλαδή θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οικολογική γεωργία να προαχθεί περισσότερο. Γιατί εκεί η εποπτεία του τι καταλήγει στις ζωοτροφές είναι μεγαλύτερη και είναι πιο ασφαλής η μέθοδη παραγωγής αυτών των ζωοτροφών. Ο Μπάς. Περιμένω μέχρι να τελειώσουν οι επιμέρους συζητήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρεμβαίνω στην συζήτηση διότι συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένα θέματα, δηλαδή με τα μέτρα που προτείνεται για την παρακολούθηση, την άμεση κοινοποίηση, διότι γνωρίζουμε ότι ήδη τα πρώτα κατάλοιπα ανεβρέθηκαν από τον προηγούμενο Μάρτιο. Νομίζω λοιπόν άμεση κοινοποίηση, άμεση επικοινωνία είναι απαραίτητη. Επίσης ε, προτείνεται μάλλον διαχωρισμό των τεχνικών λοιπόν από αυτά που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές. Μα το θέμα δεν ξέρω αν είναι αυτό. Υπάρχει νομοθεσία που τα απαγορεύει τα πράγματα αυτά. Άρα ακόμα και αν γίνει ο διαχωρισμός αυτός θα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν κίνητρα να αναμίξουν αυτά τα τεχνικά έλαια γιατί είναι φτηνότερο να τα αναμίξουν στις ζωοτροφές λοιπόν ακόμα και αν υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός, πάντοτε θα συνεχίσουν να υπάρχουν κίνητρα να χρησιμοποιηθούν με κακό τρόπο. Συμφωνώ λοιπόν με την Ντάγμαρ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι, δηλαδή να βάλουμε κάποια στοιχεία χαρακτηρισμού των τεχνικών ελαιών. Για παράδειγμα, κάποιο χρωματισμό, ώστε μόλις χρησιμοποιηθεί σε ζωοτροφή να φανεί αμέσως, αλλάζοντας το χρώμα. Αν απλώς διαχωριστούν οι δύο αλυσίδες παραγωγής, θα συνεχίσουν ωστόσο να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα θεωρήσουν ότι είναι κερδοφόρο να τα αναμίξουν. Βάλτε λοιπόν χρώμα. κυρία Γκροστέτ. Ακούστηκαν πάρα πολλά και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την τελευταία παρέμβαση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα υπάρχει και μία απάτη. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ αυστηρές, τρομερές οι κυρώσεις για να μην υπάρχουν κίνητρα να ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα σε λίγα χρόνια και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε κάποια νομικά πλαίσια έτσι ώστε να είναι αδύνατη η συγκεκριμένη επιμόλυνση της διατροφής των ζώων. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. Πρώτον, κυρώσεις, έλεγχη και ταυτόχρονα κάποιοι κανόνες, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες, κανόνες που θα εμποδίζουν αυτό το οποίο έγινε να ξαναγίνει. Ροσμπαχ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ε, επισύσω την προσοχή σε ένα πρόβλημα Βρίσκω ότι διαρκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καμιά φορά μέχρι ότου η νομοθεσία εφαρμοστεί και όλοι συμμορφωθούν. Και διαρωτώ με, τι γίνεται, πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί μέχρι ότου ένα νομοθέτημα, ένα νομοθετικό έργο, ένας νόμος πραγματικά στην Ήπεθρο στις ε, κτηνοτροφικές μονάδες εκμετάλλευσης καταλήγει και τον τηρούν αυτό τον νόμο. Είτε είναι για πουλερικά, είτε για κτηνοτροφία, είτε ηχθειοκαλλιέργειες. Εδώ υπάρχει ανησυχία για την υγεία, άσχετα το τι παράγει κανείς. Στο τέλος τέλος πάντα ταυτόχρονα είναι κανείς καταναλωτής άλλων προϊόντων. Και δεν καταλαβαίνω, δεν κατανοώ απλούστατα όταν παράγεται κάτι τέτοιο το ότι δεν υπάρχει ευθύνη από εκείνους που παράγουν κάτι τέτοιο έναντι των συμπολιτών του έναντι εκείνων που είναι δίπλα του και κοντά του, που επίσης καταναλώνουν αυγά, ψάρια και πουλερικά. Τι γίνεται με την ευθύνη αυτή δηλαδή. Και πραγματικά θα ήθελα και τα ίδια τα ζώα που έχω εγώ ε, ε, στην πατρίδα μου, τα ζώα που καταναλώνω, να μπορούμε να τα καταναλώνουμε με ίσχυ συνείδηση. Ε, souligner deux points. Le premier, c'est que je crois que vos quatre propositions vont incontestablement dans la bonne direction. οι τέσσερις προτάσει ακολουθούν μια σωστή πορεία θα έλεγα. Αλλά είπαν πολλοί συνάδελφοι και δεν μπορώ παρά να του υποστηρίξω, έχουμε ανάγκη καταρχά από την εφαρμογή των υπαρχουσών διατάξεων. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο περιορισμένων δημοσιονομικών μέσων και απελευθέρωση των αγορών. Έχει σημασία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με την πραγματικότητα των εγγράφων τα οποία ψηφίζουμε, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα το τι ψηφίζουμε. Αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, τότε δεν έχει νόημα αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο σημείο, και θα συμφωνήσω εδώ με την Φρανσουάς Γκροστέτ, οι κυρώσεις να είναι πολύ αυστηρές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία για την εφαρμογή του ποινικού περιβαλλοντικού δικαίου. Πρέπει λοιπόν να αυξηθούν οι κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθορίζει το επίπεδο των κυρώσεων, τα κράτη-μέλη το κάνουν, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι αποτρεπτικές γιατί κάθε φορά τα ίδια βιώνουμε. Και εμείς χάνουμε τρομερό χρόνο στο να νομοθετούμε εκ νέου ε, για κάποιους αποδιοπομπαίους τράγους πρέπει να βρούμε τα τεχνικά μέσα έτσι ώστε να δούμε πραγματικά ποια είναι τα επόμενα επίπεδα της διοξίνης τα οποία ε, θα επιδιώξουμε και να ελέγξουμε γενικά την κατάσταση με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι αυστηρές και ισχυρές. Και πραγματικά η νομοθεσία μας μόνο μια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη μπορεί να προβλέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί έλεγχοι και κυρώσεις. Στο τέλος τέλος όμως η ευθύνη είναι των κρατών μελών. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και να εμένουμε για αυτό το σημείο έναντι των κρατών μελών. Μετά θα ήθελα να πω δυστυχώ δυστυχώς πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε την μόλυνση με διοξίνες. Γιατί δεν είναι κάποιο περίεργο θαύμα αυτό. Ευρέως είναι παρούσα η διοξίνη διότι μολύνει το περιβάλλον ευρέως και όπου υπάρχει καύση υπάρχει παραγωγή διοξινών. Κάθε φορά που υπάρχει καύση κατοικέγεται βιομηχανικά στις βιομηχανίες. Όπου υπάρχει τέτοια βιομηχανική καύση υπάρχουν διοξίνες. Είναι έμονο αυτό το φαινόμενο, δεν αποδομείται και βρίσκεται παρόν και στα τεχνικά λύπη ε, τεχνικής μορφής έλεα πάντα εμπεριέχουν διοξίνες. Ε, αυτό που είπε η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι πιο πριν, αυτό που ανέφεραν και ενέμειναν σε αυτό, σαφώς θα συμπεριλάμβουμε αυτή την ιδέα του χρωματισμού των βιομηχανικών ελαίων. Θα τα χρωματίζουμε ώστε να μην μπορούν να αναμειγνύονται. Όμως θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όπου υπάρχει μια απάτη και σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι δεδομένη απάτη ή όχι. Συνεχίζονται οι έρευνες. Δεν ξέρουμε αν ήταν ανθρώπινο σφάλμα, αν ήταν απλώς μια ευρεία μόλυνση ή αν ήταν κάποια περίπτωση απάτης. Μπορεί να είναι και ανθρώπινο σφάλμα αυτό, ανθρώπινο λύστημα, διότι στην ίδια μονάδα έπαιρναν βιομηχανικά έλαια και έλαια από τροφές και παρήγαγαν, ξέρετε, έλαια για ζωοτροφές αλλά και έλαια για το βιοντίζερ, παραγωγή βιοντίζερ. Δεν θέλω να πω ξεκάθαρα ποιος ήταν ο λόγος ή όχι. Οι Γερμανοί είναι σοβαροί για την έρευνα που γίνεται και είπαν θα γίνει έρευνα και θα μάθουμε. Θα μάθουμε και αν υπάρχει πράγματι απάτη θα είναι αυστηρότατη η παρέμβαση. Θα πέσει πέλεκης. Αλλά αυτό το οποίο είπατε, χρωματισμός. Χρωματισμός να δούμε, να είναι με βεβαιότητα αν ήταν ανθρώπινο σφάλμα ή τι συνέβη. Για να απαντήσω όμως την ερώτηση της Ντάγμαρ. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές αναλύσεις διοξινών που γίνονται κάθε έτος, κάθε χρόνο ήθιστε συνήθως μεταξύ χιλίων και δύο χιλιάδων έλεγχοι που γίνονται για τις διοξίνες, επιτροφίμων και πολλές χιλιάδες για τις ζωοτροφές τέτοιων ελέγχων. Τι είπατε, χωρίς μικρόφωνο. Πέντε χιλιάδες, ε, πέντε είναι πολλοί έλεγχοι, δεν είναι ένας έλεγχος που γίνεται, είναι μια ολόκληρη στίβα εκθέσεων από τα κράτη-μέλη. Και όταν έχουμε ένα επίπεδο που δεν βρίσκεται ακόμα στο μέγιστο επίπεδο, αλλά πιο χαμηλά από το μέγιστο επίπεδο, επίπεδο δραστηριοποίηση όμως, action level, τότε πρέπει να κινητοποιηθούμε. Και βρέθηκε αυτό επειδή ο ε, εκμεταλλευτής, ε, ο παραγωγός ε, ζωοτροφών έκανε κάποιον έλεγχο ως ήθιστε, έναν κανονικό έλεγχο και βρέθηκε αυτή η περίπτωση, ανακαλύφθηκε. Έλεγχοι υπάρχουν λοιπόν. Τώρα, όμως, Μόλυνση φυσικά ε, σημειώνεται σε μια παραγωγή, για παράδειγμα, λοιπόν. Και κάποτε, είτε πιο πριν, πιθανότατα, γιατί υπήρχε ένας μήνας που μεσολάβησε από τη δειγματοληπτική συλλογή, από τη συλλογή των στοιχείων και μετά την ενημέρωση. Και ξεκινήσαμε, η Γερμανία ξεκίνησε, δηλαδή ε, πάγωσε την παραγωγή σε αυτή την ε, μονάδα και άρχισαν οι έρευνες. Αυτό το περιθώριο, το χρονικό δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο. Όταν υπάρχει μόλυνση πρέπει άμεσα να παρεμβαίνουμε. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε για τη, το, τη μόλυνση Κάνουμε λόγο για ένα στοιχείο μολυντικό, ένα μολυντή που υπάρχει παντού, διοξίνες. Σημαντικό είναι να το εντοπίζουμε, να τον εντοπίζουμε και να παρεμβαίνουμε άμεσα, γοργά. Το να σας εγγυηθώ δεν θα υπάρξουν άλλες τέτοιες περιπτώσεις μόλυνσης με διοξίνες είναι αδύνατο, είναι ανέφικτο. Όπως το είπα πιο πριν, πρέπει όμως να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας για την άμεση ανείχνευση και προληπτική και δραστηριοποίηση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ την Διευθύντρια της Κομισιόν. Νομίζω ότι το θέμα αυτό θα επανέλθουμε. Η Ντάγμαρ σύντομα όμως. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ό,τι είπες δίκιο έχεις. Ακριβώς όμως δεν ήταν απάντηση στην ερώτησή μου. Ξέρω ότι ο, ο παραγωγός ζωοτροφών βρήκε το πρόβλημα και αναρωτηθήκαμε ε, πόσες ποσότητες μπορεί να ελέγξει κανείς. Κατά τύχην βρήκαμε το πρόβλημα. Πράγματι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ζωοτροφές και τρόφιμα ισχύει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Γερμανία δεν γνώριζε αυτό το σύστημα, να σας το πω έτσι. Ή θεώρησαν ότι δεν ίσχυε για αυτούς. Μπορείς να θέσετε, αν θέλετε, το ερώτημα στο Υπουργείο Γεωργίας του Συμβουλίου. Ένα άλλο σημείο όμως. Ο έλεγχος των ε, τροφών και των ζωοτροφών ε, δεν ε, επιβάλλεται στα κράτη-μέλη πότε και πώς θα γίνει. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν το πότε και το πώς μα είπατε επίσης ότι τα κράτη-μέλη πράγματι ενημερώνουν για τους ελέγχους που κάνουν. Πράγματι αυτό έχει αλλάξει φαίνεται. Ενδιαφέρομαι να μάθω ε, πώς τα κράτη-μέλη αναφέρονται στους ελέγχους που έχουν κάνει και με ποιο τρόπο. Καλώς λέει κυρία Λεπάζ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι τελειώσαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν Ευχαριστώ την κυρία Ρινάλτη και τον κύριο Διευθυντή που ήρθε μαζί μας και σας προτείνω να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η παράνομη αλίευση. Ο εισηγητής μας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κυρία Ρόσμπαχ. Um, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή εδώ μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την παράνομη αλληλεία έχει αναλάβει και είναι τμήμα της νέας πολιτικής για την αλληλεία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τους αλληλείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Επιτροπή Αλληλείας λοιπόν έχουμε το πρώτο έγγραφο εργασίας ε, που τίθεται για μια, σε μια πρώτη συζήτηση την Τετάτη τώρα στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αυτό το πρώτο έγγραφο εργασίας λοιπόν που καταλήγει δεν έχει καν εγγραφή, δεν είχε καν εγγραφή στην ημερησία διάταξη στην ε, εργασία τη επιτροπή Αλίας. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα δεύτερο έγγραφο εργασία που θα μας υποβληθεί. Όμως η γνωμοδότηση φυσικά θα υποβληθεί μετά την εξέταση που θα έχει ολοκληρωθεί προηγούμενα, δηλαδή το νωρίτερο Μάρτιο ή κιόλα και Απρίλιο. Αποφασίστηκε από πλευρά τη Επιτροπή Αλία τώρα να έχουμε μια γνωμοδότηση, από πλευρά τη Επιτροπή μα να κάνουμε μια γνωμοδότηση για αυτή την έκθεση. Επικεντρώνομαι εγώ σε κάποια κύρια στοιχεία που θεωρώ ότι πρέπει να ενδυναμωθούν, να ενισχυθούν όταν πρόκειται ακριβώ για το θέμα τη καταπολέμηση τη παράνομη αλία. Για μια γνωμοδότηση όμως ε, ήταν κάτι το ιδιαίτερα χρονοβόρο και γι' αυτό προτίμησα στο κείμενο να ε, τηρηθώ σε ένα ε, γενικότερο επίπεδο. Είναι ένα έγγραφο εργασίας αυτό το κείμενο, όμως το πήρα, πρέπει να πω, την πέμπτη μόνο όταν ε, ήταν στη διάθεσή μου. Και μπορώ να δω και να πω ότι μία ολόκληρη σειρά τροπολογιών θα πρέπει να καταθέσω σε σχέση με αυτή, να κατατεθεί σε σχέση με την γνωμοδότησή μου. Έχω λοιπόν ένα πρόβλημα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα το ίδιο. Το θεωρώ παράλογο εμείς εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να συντάσσουμε μια γνωμοδότηση κιόλας και προτού η κύρια αρμόδια επί της ουσίας αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει ασχοληθεί καν με αυτό το θέμα. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς. Εμείς συντάσσουμε τροπολογίες εδώ και διατυπώνουμε ε, τροπολογίες ενώ η επί της ουσίας κοινοβουλευτική επιτροπή δεν έχει καν ολοκληρώσει. 4η Η Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, ε, για την κατάθεση τροπολογιών. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή μόλις θα έχει τότε το έγγραφο εργασία στη διάθεσή της. Αυτό είναι απόλυτα αντίστροφο από εκείνο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει μια έκθεση επί της οποίας θα πρέπει να τοποθετηθεί κανείς στην ε, συναρμόδια επιτροπή και όχι να βρίσκεται εν κενό μετέωρος κάποιος και να μην γνωρίζει επί θα τοποθετηθεί. Είναι αρνητικό αυτό όταν δεν έχουμε κάποιο έγγραφο, κάποιο στοιχείο το οποίο να μπορεί να ταιριάζει με τη, στην πραγματική έκθεση. Προσπάθησα λοιπόν εγώ κάποια ε, δευτερεύοντα θέματα να εξετάσω για τα ε, σκάφη, για την διεθνή συνεργασία, τι πρέπει να γίνει ε, μέσα στο πλαίσιο των διεθνών οργάνων και οργανισμών και συμφωνιών, τι πρέπει να γίνει, ποιος διοντολογικός κώδικας θα μπορούσε να ε, υιοθετηθεί, διότι φυσικά μεγάλο εύρος παράνομων δραστηριοτήτων, αλλιευτικών δραστηριοτήτων υπάρχει που ακολουθείτε. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι πολύ ενεργές στην παράνομη αλία, ακόμα και στο ίδιο, στην ίδια τη Μεσόγειο. Και προσπαθώ να είμαι σε επαφή με την ε, εισηγήτρια ε, Λεβίν και θα προσπαθήσω ακόμα να συζητήσω αυτό το θέμα μαζί της, σίγουρα. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι την Τετάρτη της 4 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όπως ε, προαναφέρθηκε. Επειδή θα, ναι μεν εγώ θα προσπαθήσω να αναβληθεί, να μετατεθεί αυτή η ημερομηνία, να δούμε τι θα εξεταστεί και τι θα γίνει στην Επιτροπή Αλληλείας και ποια συνέχεια θα δοθεί. Και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα με βοηθήσουν να διατυπώσω κάτι και να προτείνω κάτι το οποίο θα είναι θετικό και αποτελεσματικό και θα είναι υπεύθυνο ως πρόταση από πλευράς της ε, Επιτροπής μας διότι θα ήθελα φυσικά από την άλλη πλευρά να προστατευτεί η αλία και να προστατευτούν οι αλίες έναντι της παράνομης αλίας. Θα ήθελα να μεριμνήσουμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με προστατευόμενα, άλλες προστατευόμενες περιοχές ε, αλιές να μπορούν ε, να αλλιεύουν και θα ήθελα με αυτές τις τροπολογίες να καλύψω αυτήν την ανάγκη. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όπως είπε και η Επίτροπος Δαμανάκη, οι παράνομες δραστηριότητες στην Αλία αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και σύν της άλλης ε, ε, εισάγουμε πάρα πολλά αλλιεύματα. Ίσως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εισαγωμένων αλλιευμάτων έχουν αλλιευθεί παράνομα. Αυτό βλάπτει και το θαλάσσιο περιβάλλον και δημιουργεί και απειλές πιθανώς για το τροφιμικό περιβάλλον και φυσικά δημιουργεί προβλήματα και στις περιοχές όπου αναπτύσσονται ε, τα αλλιεύματα. Πρέπει να σταματήσει η χρήση των σημεών ευκαιρίας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι αυτές βέβαια οι οποίες υποφέρουν από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες γιατί τα αλλιεύματα για τις χώρες αυτές είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους και συνήθως αλλιευτικοί στόλοι από τις αναπτυγμένες χώρες, τις βόρειες χώρες, προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τα πιστοποιητικά για την ομιμότητα των αλλιευμάτων σε έφετο χρόνο Νομίζω ότι οι διεθνείς επιτροπές κάνουν καλά τη δουλειά τους κάπου κάπου, αλλά απαιτείται να υπάρξει μια καλύτερη αξιολόγηση και περιοδική, περιοδικός έλεγχος της αξιολόγησης αυτής. Απαιτείται επίσης λεπτομερή συνεργασία για τη συλλογή των δεδομένων από τα σκάφη και έγκαιρος εντοπισμός των σκαφών που προβαίνουν σε παράνομες αλλιεύσεις. Στίβενσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο Κρήτον και η Ρόσμπαχ. Νομίζω ότι το ότι δίνουμε μια γνωμοδότηση έχει μεγάλη σημασία εφόσον ενισχύσουμε αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή επί η Επιτροπή Αλίας και η Άννα και ο Κρήτον είπαν σωστά ότι η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα είναι τεράστια. Σε παγκόσμιο επίπεδο 10 με 23 εκατομμύρια δολάρια ο κύκλος εργασιών. Δισεκατομμύρια δολάρια λοιπόν. Uh, are Λοιπόν υπάρχουν και εδώ δυστυχώς ε, φαινόμενα μαφίας και οργανωμένου εγκλήματος, υπάρχει εκμετάλλευση και των αλλιευτικών πόρων, ιδιαίτερα στην δυτική όχθη της Αφρικής, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν παγιδευτεί να εργάζονται σε κάποια από τα σκάφη αυτά. Τους λέγεται ότι θα πληρώνονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, δουλεύουν σε απαράδεκτες συνθήκες, είδα κάποια φιλμ Αφρικανών οι οποίοι φτιαρίζουν ψάρια σε αμπάρκια χωρίς αερισμό όπου δεν μπορούν καν να σταθούν όρθιοι και δουλεύουν κάτω από τις συνθήκες αυτές 12 ώρες την ημέρα. Και πληρώνονται πραγματικά χοροϊδία είναι τα λεφτά τα οποία παίρνουν. Οι συνθήκες λοιπόν στην ουσία οδηγούν και τις συνθήκες υγιεινής αποθήκευσης των αλλιευμάτων να είναι απαράδεκτες. Πολύ συχνά τα αλλιεύματα τα οποία αλλιεύονται στην δυτική πλευρά της Σαχάρα και σε άλλες περιοχές στην ουσία περνούν στη θάλασσα σε άλλα σκάφη και πάρα πολύ συχνά φτάνουν σε λιμένες ευκαιρίες όπως τα Κανάρια από όπου παίρνουν πιστοποιητικά ότι είναι ευρωπαϊκά αλλιεύματα και ε, βρίσκουν τον δρόμο τους για τις αγορές μας. Και όπως είπε ο Κρήτον, εμείς είμαστε στον τομέα των αλλιευμάτων αυτάρκης μόνο κατά 40% και αυξάνεται η ζήτηση από το κοινό λόγω ακριβών των προβλημάτων που έχουμε με τα άλλα πρωτεϊνούχα προϊόντα όπως την βιομηχανία κρέατος λοιπά. Ακριβώς λόγω της κατάστασης αυτής ε, ο κόσμος θέλει περισσότερα ψάρια. Από πού θα προέλθουν τα ψάρια αυτά και δυστυχώς η υπεραλίευση, η παράνομη αλίευση είναι μια λύση. Δυστυχώς πολλά σκάφη ευρωπαϊκά έχουν σημαίες ευκαιρίας και οι χώρες που δίδουν τις σημαίες αυτές είναι η Ονδούρα, η, ε, ο Παναμάς και άλλες χώρες. Διαρωτώμε λοιπόν γιατί να υπάρχουν ευρωπαϊκά σκάφη με σημαίες ευκαιρίας από τις ε, χώρες αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει ένα μητρό, ε, ένα νιογνώμονας μάλλον όλων των, για όλα τα ευρωπαϊκά σκάφη και είναι σκανδαλώδες το ότι τα ευρωπαϊκά σκάφη έχουν σημαίες ευκαιρίες. Είναι σαφές ότι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες και σε εμπορία παρανόμως αλλιευμένων προϊόντων και θα πρέπει να ονοματιστούν και να εκτεθούν θα έλεγα. Συνεπώς λοιπόν η πρόταση της ΣΑΝΑ θα βοηθήσει τις προσπάθειες της Επιτροπής Αλίας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Τζαμπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην ουσία μιλάμε για ψάρια από χρυσό που δεν φυλάσσονται στο Fort Knox στις κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά στους ωκεανούς. Είδαμε τι έγινε με τον οξύριγχο, είδαμε τι γίνεται με τους ξυφίες, με τους τόνους που φτάνουν να πουλιουνται 2 2-3 χιλιάδες ευρώ το κιλό. Μιλάμε για, για χρυσάφι στη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται νομίζω έγκαιρα, έφετα η συγκεκριμένη αυτή έκθεση της Επιτροπής Αλίας και η γνωμοδότησή μας. Σε ό,τι με αφορά τώρα, εμείς η έκθεση αυτή στην ουσία θα πρέπει να καταγγείλει ένα πρόβλημα κατεπηγόντως. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Θα πρέπει να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο αδειάζουμε τις θάλασσές μας από ψάρια. Και δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε εκτός για να υπάρξει μια κάποια αλλαγή. Φυσικά υπάρχουν συνολικά προβλήματα με τις οργανώσεις, περιφερειακές οργανώσεις που δεν συμπεριφέρονται με τον σωστό τρόπο, δεν υπάρχει επιβολή των αποφάσεων οι χώρες οι αλλιευτικές δεν κάνουν ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούν την βιομηχανία τους. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα λοιπόν με την επιβολή των κανόνων και των νόμων που έχουμε. Α, πολλές φορές όμως δεν υπάρχουν κανόνες, οπότε σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα χειροτερεύει. Τι είναι, ποια είναι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γαλλικές αρχές συνεργάζονται με τη βιομηχανία τους για να νομιμοποιήσουν ε, κάποιες κατηγορίες τόνου. Ε, βλέπουμε επίσης ότι οι Ισπανοί ψηφίζουν δύο ή τρεις φορές τις ποσοστώσεις τους κατέτους και αυτό γίνεται παρανόμως φυσικά. Συνεπώς πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια αυτής της βιομηχανικής δραστηριότητας προέρχονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τα πω στην κυρία Δαμανάκη σε λίγους μήνες. Λοιπόν θα πρέπει να γίνει αυστηρότερη ακόμα η γνωμοδότηση αυτή. Ξέρω ότι η Άννα δεν είχε πάρα πολύ χώρο και χρόνο για να διατυπώσει τις πρώτες προτάσεις. Θα προσπαθήσω να τη βοηθήσω να γίνει αυστηρότερη η έκθεση. Νομίζω ότι η ενίσχυση των ελέγχων είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε έναν κανόνα πολύ θα έλεγα πιο, ένα τομέα πιο διαφανή από ό,τι σήμερα και ο Στρεμόπουλος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα που συζητούμε είναι σημαντικό και παίζονται τεράστια συμφέροντα είτε με νόμιμο είτε με παράνομο τρόπο η ανθρωπότητα έχει στραφεί σε ένα κυνήγι ζωικών πρωτεϊνών και κάνει τα πάντα για να το αποκτήσει. Υπάρχει πέρα από την καταστροφή ε, του γόνου, της δυνατότητας αναπαραγωγής. Υπάρχουν ε, τεράστιες, ε, τεράστιες βιομηχανίες που μετατρέπουν τα ψάρια σε ηχθιάλευρα, καταλήγουν στα στομάχια των κατοικίδιων ζώων και από εκεί στα πιάτα μας. Άρα χρειάζεται ένας συνολικός διαφορετικός προσανατολισμός και στον τομέα της αλίας και στον τρόπο κατανάλωσης και της διατροφής. Για να είμαστε όμως συγκεκριμένοι, θα ήθελα να εστιάσουμε σε ένα σημείο, στο σημείο 3, είναι σημαντικό να επιμείνουμε εκεί και να διευκρινίσουμε, γιατί ακριβώς αναφέρει ότι παράνομη αλία πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε διενεργείται από αλλιευτικούς στόλους τρίτων μερών, είτε από στόλους κρατών μελών. Τα καράβια με σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη βέβαια πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τον IUU ε, κανονισμό, δηλαδή αυτόν για τα παράνομα και ανεξέλεγκτα σκάφη και αυτό σημαίνει να ελέγχουν και να παραπέμπουν τα πλοία που ψαρεύουν παράνομα, να τσεκάρουν ότι τα ψάρια που εισάγουν δεν έχουν αλλιευθεί με παράνομα μέσα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες κλπ. κλπ. Ήδη από ανεπίσημες δηλώσεις ε, της τελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε καταλάβει ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να μας πει η DG Mare πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και να αποτυπώσουμε στην προσπάθειά μας και στα κείμενα τις απαντήσεις που θα πάρουμε. Ευχαριστώ. Merci infiniment. Avant de passer la parole à Sabine Wills, je voudrais... Θα ήθελα να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία α, της Σουηδικής Βουλής. Καλώς ήρθατε για να παρακολουθήσετε το τέλος της συνεδρίασής μας. Η Σαμπίν Βίλς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κάθε πέμπτο ψάρι που αλλιεύεται διεθνώς είναι παράνομο. Αυτά τα λέει η Greenpeace. Υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία ήδη από τον Ιανουάριο του 2010 κατά της παράνομης αλλιείας. Όμως η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται σχεδόν πουθενά. Διεθνώς ο τζίρος της παράνομης αλίας είναι πάνω από 10 δις ευρώ. Δηλαδή πρόκειται για πολλά λεφτά. Ιδιαίτερο πρόβλημα που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι οι σημαίες ευκαιρίας, διότι συνήθως δεν υπάρχουν περιφερειακές συμφωνίες αλίας, ούτε λαμβάνουν υπόψη οι χώρες αυτές οποιασδήποτε ποσοστώσεις αλληλευμάτων... έτσι δίνουν σε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε επιχείρηση αλίας οι χώρες αυτές ε, των ε, ε, φτηνών σημειών ευκαιρίας τη δυνατότητα να ψαρεύει οπουδήποτε. Θα προτείνω ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα να τα περιλάβει η κυρία Ρόσπαχ. Οι, δυνατότητες έχουν, οι, οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν τις, τις σημαίες ευκαιρίες, απλώς απαγορεύοντας την είσοδο των σκαφών που φέρνουν σημαίες ευκαιρίες στα λιμάνια τους. Επίσης πρέπει να απαγορευτούν οι μεταφορές των αντιευμάτων σε, χωρικά, σε διεθνή χωρικά ίδια από ε, σημαίες ευκαιρία σε πλοία άλλων σημείων. Πρέπει να διακοπεί δηλαδή το κύκλωμα αυτό από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Χρειάζεται απόλυτη ανιχνευσιμότητα. Το υπάρχει όπως είπα η νομοθεσία ίδια τον Ιανουάριο του 2010 αλλά δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή της. Η εφαρμογή της και οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να γνωρίζουν το ψάρι που αλλιεύτηκε. Όλα τα σκάφη μπορούν και πρέπει να παρακολουθούνται με τα δορυφορικά συστήματα και οι ε, αρχές επίβλεψης, εποπτείας πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά των δορυφορικών συστημάτων. Σας ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση για το θέμα αυτό. Η κυρία Μακάβαν, συγγνώμη. ακούγοντα του συναδέλφους, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Υπάρχει εδώ κάποιο εκπρόσωπος τη Κομισιόν, το γνωρίζετε αυτό κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσε ο πρόσωπος της Κομισιόν να αναφερθεί στο πρόβλημα του εύρου ε, του τζίρου της αλίας από σημαίες ευκαιρίας και οι ναυτιλιακές αρχές κλείνουν τα μάτια τους απέναντι στις παράνομες αυτές δραστηριότητες. Όλοι γνωρίζουν ότι οι ορισμένες κατηγορίες σκαφών δεν εμπίπτουν στις ε, νομοθετικές ε, ε, διατάξεις της Ένωσης και υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Πού βρίσκονται τα εμπόδια για να γίνει κάτι πραγματικά διότι εδώ και χρόνια τα συζητούμε και δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Ευχαριστώ την Άννα Ρόσπαχ για το κείμενό της, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή η νομοθεσία που υπάρχει να αρχίσει να εφαρμόζεται και να υπάρξει κάποια επίπτωση στην πράξη. Ευχαριστώ κυρία Μακάβαν. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Βερζίνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι γιατί έχουμε άλλα δύο θέματα γενικά. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε, αλλά ένα τουλάχιστον ελπίζω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που πήραν το λόγο πάνω στο θέμα αυτό που δείχνουν το επίπεδο ανησυχίας για την παράνομη αλληλεία που όλοι την λαμβάνουν υπόψη και στη δική σας Επιτροπή. Το ίδιο συμβαίνει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία βλέπει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει υπάρξει πρόοδος μετά από την υιοθέτηση από πλευρά του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων του προγράμματος το 2007 για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας και του κανονισμού ο οποίος υιοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2010, εφαρμόζεται για όλα τα αλλιεύματα, για όλες τις ναυτικές ζώνες, ανεξαρτήτως της σημαίας με την οποία κυκλοφορεί το σκάφος και ανεξαρτήτως της εθνικότητας των επιχειρηματιών και αυτό περιλαμβάνει φυσικά και τους ε, Ευρωπαίους ε, ιδιοκτήτες καφών. Βέβαια ακούστηκαν ποια είναι τα προβλήματα σε επίπεδο οργάνωσης ιδιαίτερα των περιφερειακών οργανώσεων αλίας μέσω της παρέμβασης ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών αλλιευτικών επιχειρήσεων σε μη ευρωπαϊκές ζώνες, της χρήσης των σημαίων ευκαιρίας Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία ελήφθησαν υπόψη στα πλαίσια του νέου κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός έχει σαν στόχο καθολικής εφαρμογής, σχεδόν καθολικής, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δεσμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί που υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι ο κανονισμός αυτός, ο οποίος έγινε δεκτός ανταποκρινόμενη στις ελλείψεις που υπήρχαν δεν θα λειτουργήσει πλήρως παρά μόνον αν και άλλες ε, εμπλεκόμενες πλευρές συνειδητοποιήσουν το κατεπήγον του προβλήματος και καταπολεμήσουν την παράνομη αλία, εμπνευστούν από τα συστήματα τα οποία έχουν τεθεί ε, σε λειτουργία στην Ένωση έτσι ώστε να υπάρξει ένα θα έλεγα δυσόπιτο κυνήγι των παρανόμων ε, αλλιευτών. Είχαμε κάποιες βελτιώσεις ε, μέσα στον πρώτο χρόνο του κανονισμού αυτού. Είδαμε ποιες είναι οι τεράστιες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε λόγω της αντίθεσης ορισμένων τρίτων χωρών. Είδαμε επίσης και μια κάποια αντίσταση σε εισαγωγικά από πλευρά των ε, επιχειρηματικών κύκλων και των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών αλλιευτικών κύκλων. Γι' αυτό λοιπόν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της νέας συνθήκης ενός ε, νέου μέσου θα έλεγα συντονιστικού και θα απαιτήσει οι κυρώσεις ε, να εφαρμοστούν πλήρως. Ταυτόχρονα όμως ε, δεν θα είναι χρήσιμα τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας παρά μόνο εάν σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο ΕΦΑΟ και σε επίπεδο όλων των οργανώσεων των περιφερειακών των Ηνωμένων Εθνών, των αλλιευτικών περιφερειακών οργανώσεων και όλων των εμπλεκομένων χωρών που προσφέρουν τη σημαία τους ή εμπορεύονται τα προϊόντα αυτά, τα μέτρα αυτά εφαρμοστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σας ευχαριστώ κύριε Βερίν. Κυρία Ρόσμπαχ, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών θα παραταθεί. Κανονικά θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση στις 17 Μαρτίου και στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Αλλά θα δούμε ίσως αν υπάρξει μια μετάθεση χρονική όλων αυτών των ημερομηνιών. Καλώς. Περνάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο τελευταίο. Η κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ. Θέλω τώρα ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση να πούμε, να δύο λόγια. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν καλά αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να το δω αυτό ακριβέστερα προτού το πιστέψω. Να το δω πιο εξειδικευμένα. Στην Δανία όμως έχουμε θετικά καλά αποτελέσματα τα οποία σημειώθηκαν σε σχέση με εκείνους τους αλληλείς που αλλιεύουν έντιμα. Έντιμα. Διότι εκείνοι χρησιμοποιούν ένα GPS ε, στις στράτες τους, ώστε να μπορεί κανείς να εντοπίζει πού αλλιεύουν ακριβώς. Συζήτησα με αρκετούς αλείς και μου είπαν πολύ καλή αυτή η ιδέα, πολύ καλό. Διότι κανείς δεν μπορεί να έρθει και να πει μετά και να πει εμείς ψαρεύουμε παράνομα. Βλέπετε, ευχαρίστως ακολουθούν αυτή την πρόταση και αυτό θα μπορούσε να ήταν μια λύση μελλοντικά. Πέρα από αυτό, αληθεύει βέβαια αυτό, όπως ακούω, και κάτι άλλο, ότι εδώ αλλιεύεται χρυσός εντός εισαγωγικών. Είναι χρυσές αυτές, χρυσοφόρες αυτές οι δραστηριότητες. <laughs> Και τα παράνομα αλλιεύματα, τα παράνομα ψάρια, όχι μόνο ε, τα μεταποιούν σε ηχθιάλευρα, τίποτα δεν πετάγεται δηλαδή, κανένα ε, ψάρι δεν ε, ε, πετάγεται χρησιμοποιούνται ακόμα και για την ε, παραγωγή ηχθιαλεύρων. Όμως οι ξηφίες και ο θήνος, ο τόνος είναι χρυσά αλλιεύματα και αυτά είναι εκείνα τα οποία αλλιεύονται παράνομα πολύ συχνά. Και όλο και περισσότερο αυτές οι τράτες, αυτές οι τράτες είναι μεγάλες, είναι τεράστιες και είναι τόσο ακριβές για αυτούς αλλιείς, για τους ψαράδες που τεράστιες ποσότητες ψαριών πρέπει να συλλέγονται, να αλλιεύονται παραπάνω από τις ποσοστώσεις τους ώστε να αποσβεστεί η τιμή αγοράς τέτοιων τεράστιων σκαφών. Και όταν έχουν ε, τραβήξει τα δίχτυα στο κατάστρωμα, είναι στην κουβέρτα, είναι ε, τελείως αδιάφορο το ποιο είναι το μάτι, το μέγεθος των ματιών των δίχτυων. Ό,τι έχει ψαρευτεί χρησιμοποιείται, διότι αν, ε, όταν συλλέγονται τα δίχτυα, κάθε ψάρι είναι εκείνο το οποίο καταλήγει στα μπάρια, στα ψυγεία. <laughs> δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να ζουν σε αυτά τα δίκτυα, αυτά τα ψάρια, α, ακόμα και αν το, τα μάτια των δικτυών επέτρεπαν να ε, εξέλθουν αυτά τα ψάρια. Και έτσι πρέπει λοιπόν έτσι να προστατευτούν οι έντιμοι, οι ακέραιοι αλληλείς. Και είναι ένα σκάνδαλο, είναι σκανδαλώδες ότι υπάρχει τέτοιο εύρος παράνομης αλληλείας. Ε, ε το πω έτσι, τελείωσα εκτός κανόνων και διατάξεων αλληλείας. Ελπίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να υιοθετηθούν τέτοια μέτρα και ότι πρέπει να υιοθετηθούν και κυρώσεις για εκείνους που συλλαμβάνονται να αλλιεύουν παράνομο. Euh, είμαστε πολλοί εμείς που θα υποστηρίξουμε το αίτημά σας. Απόλυτα θεμητό αίτημα. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε ποσοστώσεις από τη μία και από την άλλη ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει είναι απαράδεκτο και αβίωτο για τους αλληλείς οι οποίοι θέλουν να είναι νόμιμοι. Καλώς. Τώρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της νομοδότησής μας για τον οικονομικό της κανονισμό της ολοκληρωμένης αλληλευτικής πολιτικής. Γνωμοδότηση για την Επιτροπή Τράνη, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας. Είμαι συγγήτρια και γι' αυτό θα σας δώσω σύντομα το περιεχόμενο της νομοδότησης αυτής και μπορεί να γίνει συζήτηση στον λίγο χρόνο που θα έχουμε. Γιατί ο κανονισμός αυτός και γιατί σας προτείνω να τον υποστηρίξουμε. Μέχρι τώρα η χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ολοκληρωμένης αλληλευτικής πολιτικής δεν έχει τύχει αντικείμενο εγγύησεων. Δεν βασίζεται παρά μόνο στις προβλέψεις του δημοσιονομικού κανονισμού που προβλέπει δύο πράγματα. Πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι βιώσιμη η πρόταση αυτή λοιπόν και ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικό δύσκολο απειλείται η ίδια η επιβίωση της ολοκληρωμένης αλληλευτικής πολιτικής που δεν θα έχει δημοσιονομικά μέσα για τις υπόλοιπες ε, δημοσιονομικές προοπτικές 11-13. Συνεπώς η Επιτροπή προτείνει τον κανονισμό αυτό και θα πρέπει να εκφράσουμε νομίζω τη στήριξή μας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μετριοπαθής, ολίγα εκατομμύρια για δύο χρόνια βέβαια και νομίζω ότι στο παρόν πλαίσιο είναι πολύ λογικό εφόσον δεχθούμε ότι αυτό είναι ένα όριο το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβούμε. Γιατί αν το υπερβούμε νομίζω δεν θα έχουμε τίποτα πλέον δημοσιονομικά στη διάθεσή μας, κανένα περιθώριο. Πρόκειται για μια έλογη πρόταση στο σημερινό πλαίσιο η οποία δεν θα πρέπει όμως να μειωθεί το ποσό το οποίο προτείνεται. Στη γνωμοδότηση την οποία προτείνω Υπάρχουν προγράμματα που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, την νεότητα και θα πρέπει επίσης ε, να βελτιωθούν τα προγράμματα για όλους τους νέους σε σχολικό και πανεπιστημιακό επίπεδο. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, αλλά και σε άλλα επίπεδα χαμηλότερα. Προτείνω επίσης να διευκρινιστούν οι στόχοι του προγράμματος. Ανάμεσα στους γενικούς στόχους έχουμε την προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης, της αηφόρου εκμετάλλευσης των αλλιευτικών και παρακτήων πόρων και της ανάπτυξης των στρατηγικών ανά θα έλεγα αναλιευτική περιοχή, όπως ακριβώς το κάνουμε και σε επίπεδο των εσωτερικών υδάτων. Προτείνω επίσης να διευκρινιστούν οι ειδικοί στόχοι και τελευταίο σημείο είναι η επιτροπολογία. Δεν άπτεται τη έκθεσή μου, αλλά υπάρχει μια τροπολογία για το πολιετές πρόγραμμα εργασία το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 7 του κανονισμού. Αυτή τη στιγμή υιοθετηθούν τα προγράμματα, καθορίζονται οι συγκεκριμένες προτεραιότητες. Διαρωτώ λοιπόν, αν η νέα διαδικασία εξέτασης, η μη διαβουλευτική, είναι χρήσιμη. Νομίζω ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει και να κρατήσουμε τις αρμοδιότητές μας και να διασφαλίσουμε τη συνοχή των πρωτοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και των εθνικών κρατών μελών από την άλλη. Θα τα συζητήσω τα θέματα αυτά επί της ουσίας με τον αρμόδιο εισηγητή τον κύριο Κουμουτσάκο. Να προσθέσω εδώ ότι ήδη συζητήθηκα με τον κύριο Κουμουτσάκο, δεν συζητήσαμε το τελευταίο θέμα όμως, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτά είχα να πω πάρα πολύ σύντομα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Στην διάθεσή μας δυστυχώς. Αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα βοηθήσει την επιβίωση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για την θαλάσσια πολιτική, θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μετριοπαθής, αλλά είναι σε βάθος, πάει σε βάθος, εμπεριέχει τα σωστά αναγκαία πράγματα. Καταρχήν, πρέπει να μιλήσουμε σε σχέση με την έρευνα, τι γίνεται. Διότι συμφωνούμε ότι η κατάσταση στις θάλασσες ε, παγκόσμια επιδεινώνεται και είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε, να υποπτεύσουμε το τι συμβαίνει και να το παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς. Το χαιρετίζω σε σχέση με το ότι ε, για τις τροπολογίες ε, αναφέρονται πράγματα όπως τα θέματα της έρευνας και η ενεργειακή πολιτική, η ενέργεια που αποκομίζουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από σε σχέση με τις απομακρυσμένες περιοχές και όλα τα σχετικά και θα έλεγα όταν πρόκειται για τα θέματα μόλυνσης και ρήπανσης επικεντρώνεται κανείς στις ε, μεταφορές ε, και στην άντληση πετρελαίου. Θα έπρεπε όμως ε, και για άλλες προβληματικές τέτοιες αιτίες να γίνεται λόγος. Επίσης, περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε σχέση με τρίτες χώρες είναι σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι θέλουμε να αποστείλουμε το μήνυμα ότι και οι τρίτες χώρες όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι τρίτες χώρες ε, πρέπει από κοινού να επομισθούν ε, δεσμεύσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, από κοινού με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ακαθόδες ε, θέμα, φλέγον θέμα. Θα ήταν ευκταίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει το δυνατόν πιο γοργά να συμφωνήσει τι πρέπει να γίνει. Επιπλέον θα πρέπει οι ευάλωτες ζώνες και ευαίσθητες περιοχές, περιοχές των ζωνών Natura, του δικτύου Natura 2000, για την προστασία της φύσης 2000 η βιοπικιλότητα σε αυτές τις ζώνες να υποστηριχθεί και να προστατευτεί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να φανταστεί κανείς ότι δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία σχετικά με την ολοκληρωμένη αντίληψη για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Η πρότασή σας, ε, κυρία Λεπάλ, είναι πόσο μου φαίνεται σωστή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες πιστώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στο περισσόριο του προϋπολογισμού για την αλλιευτική πολιτική. Αυτό ε, δεν σημαίνει πολλά πράγματα γιατί τα ποσά αυτά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη, να καταλάβουμε ότι η δραστηριότητα αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία και να διαθέσουμε περισσότερες πιστώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι ως εισηγήτρια του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής μας κάνετε μια φιλότιμη προσπάθεια να ενσωματώσετε την περιβαλλοντική διάσταση. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση της Επιτροπής απέχει κατά πολύ από το να θεωρηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση η ανεπαρκέστατη αναφορά σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και στο ρόλο που καλείται να παίξει η ναυτιλία στην αντιμετώπιση τους θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην προστασία των οικοσυστημάτων και την ορθή διαχείρισή τους. Θα θέλαμε να δούμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, ιδίως ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνδυασμένες μεταφορές, για παράδειγμα, ή τη μετάβαση από τις ε, χερσαίες θαλάσσιες μεταφορές, ε, από τις χερσαίες τις θαλάσσιες μεταφορές ή τη σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών, για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές. Προφανώς μας ενδιαφέρει το πόσα, αλλά και το πού θα διατεθούν τα χρήματα. Θα θέλαμε να δούμε καλύτερη χρήση των κονδυλίων από το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, αλλά και να υπάρξει μεγαλύτερη μέρημνα στο σχεδιασμό των παράκτιων εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κλιματικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να τονιστεί επιπλέον περισσότερο ο χωρικός σχεδιασμός ότι θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προσέγγιση των ε, οικοσυστημάτων, να ενσωματώσει περισσότερο τους στόχους της περιβαλλοντικής ομοθεσίας κυρίως για την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων, την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, την οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και την οδηγία πλαίσιο για το νερό. Επίσης, για την αντιμετώπιση της ρήπανσης από χερσαίες πηγές, πρέπει να βρεθούν οι διασυνδέσεις με την κοινή αγροτική πολιτική που συζητιέται αυτή τη στιγμή το άμεσο μέλλον της και επιπλέον χρειάζεται μια πιο εκτενής αναφορά και διασύνδεση με την κοινή αλλιευτική πολιτική. Πρέπει να ενσωματωθούν στο χωρικό σχεδιασμό καλές πρακτικές, αλλά και να γίνει εκτεταμένη χρήση των τεχνικών εκτίμησης επιπτώσεων στο παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον. Και τέλος, θα πρέπει να ενσωματωθεί η προσέγγιση του καθαρού πλοίου, γιατί η μεγαλύτερη ασφάλεια της νασιπλοείας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Euh, Εσείς κύριε Στίβενσον. Oui, Monsieur Stevenson. Vous n'avez pas demandé la parole Α, δεν έχετε ζητήσει το λόγο. Καλά. Η κυρία Βίλς. Ναι, Ευχαριστώ κυρία Λεπάζ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει για την ε, προστασία των θαλασσών. Η ποικιλότητα των θαλασσών πρέπει να, διατηρηθεί ώστε να διατηρηθεί και ο χαρακτήρας ε, ως ε, πλουτοφόρου περιοχής ο, η θάλασσα, της θάλασσας. Και εδώ εντάσσεται βέβαια και η προστασία από, την, ε, από τοξικές και από θείο. Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας στις παράκτητες περιοχές, για παράδειγμα τουρισμός και αλία. Δεν υπάρχουν ωστόσο μέτρα πρακτικής εφαρμογής κατά της υπεραλίευσης, δηλαδή εξασφάλιση για παράδειγμα ε, βιοτόπων για τα ψάρια. Επίσης παρακολούθηση και ανιχνευσιμότητα στον τομέα της αλίας που πρέπει να βελτιωθούν ώστε να αποφεύγεται η παράνομη αλία. Και επίσης πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των ε, παραλιευμάτων που ξαναπεταγόνται στη θάλασσα. Η νομοθεσία δεν είναι ισορροπημένη. Τονίζεται πολύ περισσότερο η χρήση από την προστασία. Έχω την εντύπωση ότι η προστασία αναφέρεται μοναχά όπου αποτελεί προϋπόθεση για βελτιστοποίηση ή για μεγιστοποίηση της ωφέλειας, ενώ χρειάζεται μια πολυσχηδής και πολυδιάστατη προστασία. Περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον ναυσιπλοεία, προστασία των ωκεανών και περιορισμός της παράνομης αδείας. Η κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ πολύ, Κορίν. Πραγματικά πολύ καλή δουλειά είναι αυτή, αυτή που έκανες. Συμφωνώ και με τον Έλληνα συνάδελφο ότι πραγματικά το θαλάσσιο περιβάλλον και το χερσαίο περιβάλλον συνδέονται, αλληλοσυνδέονται και μάλιστα πολύ στενά το ένα με το άλλο. Πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά είναι μια ενότητα, μια ενότητα που δεν μπορούμε να κατατμήσουμε ή να να χωρίσουμε εμείς. Ερώτηση, τι γίνεται σε σχέση με τον επιμερισμό ευθυνών ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιμέρους κρατών, των δήμων και κοινοτήτων σε σχέση με τις χώρες μας. Ποιος επομίζεται ποιες ευθύνες, ποιος είναι για ποιο θέμα αρμόδιος ως υπεύθυνο. Μπορεί κανείς, κάποιος να απαντήσει, ίσως η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Anna, euh, Madame Benini pour la Commission. για την κυρία Μπενίνη. Chairman. Thank you, Madam Chairman. Uh, First of all, we are, the Commission is very grateful for the speed in which uh, this committee has drafted this opinion. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την uh, γνωμοδότησή σας. Είναι μείζον το πολιτικό θέμα. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια νομοθετική πρόταση μετά από δύο-τρία χρόνια προπαρασκευαστικών δράσεων και απαιτείται η πλήρης υποστήριξή σας αν πρόκειται να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια διατομιακή θα έλεγα προσπάθεια. Εμείς δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε υπάρχουσες πολιτικές, θέλουμε σε αυτές τις τομεακές πολιτικές να προσθέσουμε αξία, διασφαλίζοντας συνέργειες, συνδέσμους και αηφορία στις πολιτικές αυτές, εφόσον αφορούν φυσικά την θάλασσα στην οποία θα έλεγα εξελίσσονται. Και αυτό μας οδηγεί στις δράσεις τις οποίες προτείνουμε, τη συνέχιση της χρηματοδότησης τα τελευταία δύο χρόνια των μέσω των προοπτικών, δράσεις οι οποίες στην ουσία συνεχίζουν αυτό το οποίο έχουμε κάνει, αυξάνουμε τις γνώσεις μας, αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε είναι όπως είπατε οι προτάσεις αυτές ε, μετριοπαθεί σε επίπεδο ποσοτικό, είμαστε στην αρχή, είμαστε σε επίπεδο ελέγχων, ενημέρωσης, σεμιναρίων, συγκέντρωσης πληροφοριών και με κάποια θα έλεγα μέσα τα οποία πρώτον ελέγχουν την κατάσταση της θάλασσας ποιες είναι οι δράσεις δηλαδή που μπορεί να γίνουν. Δεύτερον, τον προγραμματισμό, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σχετικά με την βέλτιστη χρήση του θαλασσίου χώρου. Και τρίτον, με ποιο τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητες που ε, εξελίσσονται στη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας. Μία παρατήρηση μόνο. Οι προτάσεις τις οποίες κάνετε σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αν και δεν διευκρινίζονται συγκεκριμένα στα πλαίσια της υπάρχουσας πρότασης γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους, απασχόληση και συνολικές δράσεις κατάρτισης έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την δραστηριότητα που επιθυμούμε. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους. Όπως βλέπετε φτάσαμε 6.30, δυστυχώς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κρίμα, γιατί τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολύ ενδιαφέροντα. Παρ' όλα αυτά είναι 6 και έχουμε ουσιαστικά εξαντλήσει ε, την ημερήσια διάταξη. Ήταν πολύ πυκνή η ημερησία διάταξη και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τελευταίο θέμα. Παρουσιάζω συλλογικά, συγγνώμη, στους συναδέλφους και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήρθαν για αυτό το θέμα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για τη συνέχεια των